Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να καθίσετε. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Σημείο 1 και έγκριση της ημερησίας διατάξεως καταρχάς. Θα ήθελα να επισημάνω το σημείο 10 που αφορά την εξέταση των τροπολογιών της κυρίας Δεκάστηλ για την ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό, καθώς και το σημείο 20 την με την εξέταση των τροπολογιών της εκθέσεως Μπάουερ για τη θέση του φίλου στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εθνικών Στρατηγικών Στέδαξης των Ρωμά, θα αλλάξουν θέση. Θα αντιστραφούν. Σημείο 19 έκθεση του κυρίου Μπουλόν και εξέταση των τροπολογιών. Θα το δούμε σήμερα το πρωί, πριν από το σημείο 11. Και αν δεν έχετε αντιρρήσεις... Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Τώρα στις ανακοινώσεις. Έκθεση ΑΦΚΟ, τροποποίηση του άρθρου 81 του κανονισμού διαδικασία έγκρισης όπως ονομάζεται. Κατόπιν ε, των συζητήσεων στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών, οι συντονιστές για την ε, Επιτροπή Απασχόλησης ε, Απεφάσισαν να εκδώσει γνωμοδότηση η Επιτροπή μας με τη μορφή της τροπολογίας, τροποποίησης στην έκθεση της Επιτροπής ΑΦΚΟΝ, σταγματικών υποθέσεων. Προβλέπεται έως τις 19 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα η κατάθεση τροπολογιών για να γίνει συζήτηση στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίασή μας. Σας υπενθυμίζω ότι η διαδικασία αυτή επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει τυπώνει ε, γνώμη, σύμφωνη γνώμη σε κάθε διαδικασία διεθνών συμβάσεων και όταν υπάρχει κάποια εταιρική σχέση με μία χώρα για θέματα απασχόλησης, εάν περάσει το άρθρο 1 όπως το έχει συντάξει τώρα η Επιτροπή ΑΦΚΟ, οι νομοθετικές επιτροπές δεν θα μπορούν να προβάλλουν τις γνωμοδοτήσεις τους, θα εξαφανίζονται δηλαδή αυτές. Ε, γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους συναδέλφους, συντονιστές, επιτροπές, πολιτικά κόμματα να προσέξουν πάρα πολύ αυτή την ε, έκθεση Ρατσκόφης και επαναλαμβάνω τροποποίηση του άρθρου 81. Δεύτερον, στα σιδηροδρομικά έχουμε αποφασίσει ο κύριος Νταγντέν ε, που έχει αναλάβει την έκθεση να ε, διατυπωθεί γνωμοδότηση για τις τρεις πτυχές της, Επιτροπή, της εκθέσεως ε, με, στην Επιτροπή Μεταφορών του κ. Νταγδέν, γνωμοδοτήσεις λοιπόν για, τους, για τις τρεις πτυχές, αλλά όχι γνωμοδότηση για τον κανονισμό 1192 καθώς 69 για τους ισολογισμούς των στυλοδρομικών επιχειρήσεων. Ο εισηγητής άλλωστε μας επεσήμανε ότι για το θέμα αυτό δεν φαίνεται σκόπιμη η ε, παρέμβαση με γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Απασχόληση. Τρίτη ανακοίνωση. Ε, έκτακτη συνεδρία των μέλων της Επιτροπής μας στις 10 Οκτωβρίου προβλέπεται προκειμένου να συζητηθούν, να θυγούν και να καλυφθούν τα καταπήγοντα ζητήματα που μα περιμένουν εν ώψη τη ολοκλήρωση της θητεία. Ε, Πέμπτη πρωί και πάλι αυτή η συνεδρίαση για την, ε, τους πόρους διερμηνίας που έχουν ζητηθεί αλλά δεν αξιοποιούνται. Με λύπη μου σας ενημερώνω ότι εχθές το βράδυ η γαλλική και αγγλική διερμηνία που είχε προβλεφθεί για τέσσερις ώρες για τον τριμερή διάλογο για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν αξιοποιήθηκε. Ο Φρέντρικ Ταρντέν δεν μπόρεσε να παραστεί στην συνεδρίαση αυτή. Σημείο 5 των ανακοινώσεων. Καλά, έχετε σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έγγραφα. Ξέρετε ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίαση από το διαδίκτυο και έχουμε πλήρη διαφάνεια εργασιών με βάση και τους προσανατολισμούς μας όσον αφορά αυτά τα θέματα. Στο σημείο 3 θα παρακαλέσω την Βερονίκα Λόπε Φοντανή να μας παρουσιάσει τις 17 συμβαστικέ τροπολογίες για την έκθεσή της για το ε, εξάμεινο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Στονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, εφαρμογή των προτεραιότητων για το 2013, πρόκειται για γνωμοδότηση για την Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο. Έχω πράγματι 17 συμβαστικέ τροπολογίε που ουσιαστικά τι τροπολογίε που παρουσιάστηκαν. Στι συμβαστικέ τροπολογίε φτάσαμε σε κάποιε ε, ε, συνεννοήσεις ε, για το πώς θα πετυχούμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Επίσης υπάρχει και άλλη συμβαστική τροπολογία για την ευελιξία της εργασιακής αγοράς με υψηλά πρότυπα κοινωνική προστασίας, μεταρρυθμίσεις εργασιακές, που βελτιώνουν την κατάσταση των ευπαθών ομάδων, μειώνουν την ανέχεια στην εργασία και συμφιλιώνουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Και επίσης ε, καταλήξαμε σε συμβιβασμό για να μειώσουμε την φορολόγηση και ε, να αυξήσουμε την περιβαλλοντική φορολόγηση. Επίσης, να βελτιώσουμε την προσληψιμότητα των νέων και επικεντρωθήκαμε ε, στην ε, έβρεση εργασίας, ε, στην απασχολησιμότητα των νέων, κυρίως όσων βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση, επίσης πρόσβαση ποιότητας και κυρίως όταν υπάρχουν καταστάσεις κρίσης. Επίσης, άρση των εμποδίων στην ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων για να έχουμε βελτίωση της κινητικότητας. Πάντοτε λέγαμε ότι θέλουμε να έχουμε κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά με εκούσιο χαρακτήρα και κατόπιν αναγκαιότητα μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τονίζοντας και τη συμμετοχή των συνδικάτων και των εθνικών κοινοβουλίων. Θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά στο συμβιβασμό ΕΛ, που όταν το συζητήσαμε με τους σκιώδεις το Άλντε είχε ζητήσει να αντικατασταθεί ο όρος κατάλληλη ε, αποζημίωση με τον όρο κατάλληλη χρηματοδότηση. Το δέχτηκε ο συγκητής έτσι λοιπόν, αντί για τη χρηματοδότηση διατηρήσαμε τον όρο αποζημίωση. Εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους φιλελευθέρους και ελπίζω οι φιλελεύθεροι να υπερψηφίσουν. Αυτά κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκαναν ε, πολύ σημαντική δουλειά. Μάλιστα και μέχρι χθε το βράδυ προσπαθούσαμε ε, να τελειοποιήσουμε όλες τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, merci, Σας ευχαριστώ. Ο Σπρέτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την εισηγήτρια για το έργο της για τη δουλειά της αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες προσπαθήσαμε τα μάλλα για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ικανοποιητική, σε κάποιους συμβιβασμούς που να μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε πλήρως την έκθεση. Και εγώ νομίζω ότι και οι περισσότεροι συμβασμοί ικανοποιούν και τη σοσιαλιστική ομάδα. Είναι αλήθεια ότι εμάς θα μας άρεσε να πάμε πιο μακριά σε ορισμένα ζητήματα που πιστεύουμε ότι έμειναν κάπως μητελή, κυρίως όταν μιλάμε ε, για την ε, δημοσιονομική εξυγίανση και βλέπετε τι βιώνουμε σε ορισμένες ε, χώρες. Το απλό ε, να ζητήσουμε, όπως ζητάει η συμβαστική τροπολογία, μία αναθεώρηση. Νομίζω ότι είναι μία θετική πρόοδος, όμως επίσης μας ε, ανησυχεί που εμείς από την Επιτροπή Επασχόλησης φαίνεται να είμαστε οι τελευταίοι ε, που λέμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμη ε, και το Διεθνές Νομοσμητικό Ταμείο έχει αναγνωρίσει ότι έχει ε, ουσιαστικά αυτή η δημοσιονομική συγκίνηση προκαλέσει μεγάλη αδικία και μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να κάνουμε και κάποια αναφορά σε ό,τι αφορά την αλλαγή της δημοσιονομικής εξυγένσης σε διορθωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί εκεί μπορούμε να έχουμε αρνητικές συνέπειες και σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά θα μπορούσε να ζημιώσει σημαντικά και το κράτο πρόνοιας και κυρίως αν ε, και συμφωνώ με τους ε, συμβιβασμούς, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε διάφορες τροπολογίες που υπάρχουν στην έκθεση και αναφέρεται στον κοινωνικό πυλώνα, στην κοινωνική ένωση και σε αυτή την ε, στρατηγική την κοινωνική. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες της κυρίας Προέδρου και κάποιες δικές μου τροπολογίες που αναφέρονται όχι στο μοντέλο κοινωνικών δικτών ε, και ε, αυτόματης σταθεροποίησης που θέλουμε να εισαγάγουμε στην ΟΝΕ, απλώς κάνουμε μία έκκληση στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτυχθεί μια πράσινη βιβλός, για να έχουμε αυτούς τους σταθεροποιητές και να συζητήσει το Κοινοβούλιο επ' αυτόν και δεύτερον να σεβαστεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει, κάτι που έκανε η Κομισιόν στο Blueprint πέρσι το Δεκέμβριο, να παρουσιάσει άπαξ μια πρόταση για το ζήτημα αυτό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο και δεν κατανοούμε γιατί κάποιες πολιτικές ομάδες έχουν αμφιβολίες για αυτές τις τροπολογίες, γιατί σίγουρα έχουν συζητηθεί αυτές οι τροπολογίες, έχουν εγκριθεί στην Επιτροπή και μάλιστα με βρει υποστήριξη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου πριν λίγους μήνες. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θέση αυτή, γιατί αναμφισβήτητα θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει έτσι πιο κοινωνική και πιο δίκαιη και θα απαντήσει και στις ανησυχίες των πολιτών. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια για το έργο της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Εάν όχι, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο Σέρχιο Κουτιέρεθ. Εξετάζουμε το ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης. Για μας είναι ένα ραντεβού πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται η κοινωνική και η οικονομική πολιτική και πώς θα λαμβάνει αυτή η υπόψη τις προτεραιότητές μας. Είναι η τρίτη φορά που το κάνουμε. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κώδικες και στα πλαίσια αυτά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και πρακτική διάσταση που είναι η εξέταση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε κράτος μέλος και μετά υπάρχει και ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι κοινωνικές και κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος θα εξετάσουμε την, εξετάζουμε την έκθεση της Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ την στιγμή που η Κομισιόν θα δημοσιεύσει επιτέλους την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Την κατάσταση δηλαδή που επικρατεί. Και αν θέλουμε και εμείς να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση αυτή, ε, με την κοινωνική διάσταση δηλαδή της ΟΝΕ, θα πρέπει να δώσουμε κι εμείς ποια είναι τα διδάγματα τα οποία έχουμε εξάγει από την, ε, τις ε, μελέτες που κάνουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια συζήτηση και όσον αφορά τους δείκτες, αλλά και να δούμε την δυνατότητα να εξερευνήσουμε, αν θέλετε, ε, την, περίπτωση να υπάρχει μια ελάχιστη ευρω... Ε, ε, ε, αποζημίωση ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να επωφεληθούμε και από την έκθεση της Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ για να ενισχύσουμε το μήνυμά μας. Ούτω ή άλλω πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και τον επόμενο μήνα, όταν συζητάμε την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα πάνω στο οποίο συμφώνησαν οι συντονιστές ή θα συμφωνήσουν οι συντονιστές μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν. Πιστεύω ότι ε, ένα μήνυμα της δικής μας ε, Επιτροπής, πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της, θα ήταν απόλυτα λογική. Ξέρω βέβαια ότι ορισμένες πολιτικές ομάδες διαρωτώνται ακόμα, υπάρχουν ε, πλανώνται ερωτηματικά, αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε τη συνεισφορά της δικής μας Επιτροπής ε, σε αυτό το θέμα και να περιοριστούμε μόνο σε αυτά τα οποία λέει η Οικονομική Επιτροπή. Εκείνοι ξέρω ότι δεν θέλουν να η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δεν θέλουν να μιλάμε για δείκτες. Δικό τους το πρόβλημα όμως αυτό. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε την σωστή όθηση προς την σωστή κατεύθυνση. Εάν δεν υπάρχει κανένα άλλο που ζητάει το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, δεν μπορώ να προσθέσω πολλά. Ελπίζω να έχει καλή έκβαση αυτή η γνωμοδότηση και να εγκριθεί στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Γιατί συμφωνώ με την Πρόεδρο, είναι σημαντικό και η φωνή της της Επιτροπής Απασχόλησης να ακουστεί και να μπορούμε να προωθήσουμε αυτά που πιστεύουμε. Πάντοτε υπάρχουν αποκλήσεις και είναι δύσκολο όχι μόνο να φτάνουμε σε συμφωνίες μεταξύ κομμάτων αλλά και εντός των ίδιων ομάδων μεταξύ των κρατών, μεταξύ των συνισωστών που εκπροσωπούν διαφορετικά κρατημέλη. Μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορές λοιπόν, αλλά πρέπει να καταλήγουμε σε συμφωνίες. Ελπίζω λοιπόν εγώ να προωθηθεί καταλήλως η γνωμοδότηση και τελικά να αντικατοπτρίζει τα όσα θέλουν όλοι οι βουλευτές αυτού του κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε επομένω σε λίγο. Και το κείμενο θα εξεταστεί από την ε, Οικονομική Επιτροπή 30 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώσαμε με το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και θα δώσουμε το λόγο στον Άνταμ Κόζα για το θέμα της, των γυναικών με αναπηρία. Είναι μια έκθεση με πρωτοβουλία της ε, Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Κυρία Κόζα, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πιστεύω ότι πρόκειται για μία... Πιστεύω ότι πρόκειται για μία έκθεση, λέει ο κύριος Κόζα, που στο που την χάνει της υποστήριξης όλων των ε, επιτροπών και όλων των ομάδων ε, και ε, όσον αφορά το περιεχόμενο. Έχω, έχουν υποβληθεί 38 τροπολογίες, εκ των οποίων οι 33 καλύφθηκαν από συμβαστικές τροπολογίες. Εκτός από δύο-τρεις τροπολογίες πιστεύω ότι οι συμβαστικές θα τύχουν υπό τις υποστήριξεις των άλλων. Όμως υπάρχουν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που δημιουργούν πρόβλημα και υπάρχουν κάποιες... Ε, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε κάθε περίπτωση ή να, υπογρα... να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε την δυσμενή κατάσταση στην οποία, δυσμενή θέση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες με αναπηρία και να τονίσουμε τη δράση που πρέπει να αναλυφθεί για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Το Z και AS οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες, είναι τροπολογίες που κατά την άποψή μου αντικατοπτρίζουν μια πολύ, ένα πολύ σαφή προσανατολισμό όσον αφορά την ε, στάση της Επιτροπής Γυναικών, τις θέσεις στην Επιτροπή Γυναικών. Έχω προετοιμάσει αρκετές ε, εκθέσεις στο παρελθόν, πρέπει να σας πω, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι η έκθεση της ε, Επιτροπή της κατουσίαν αρμόδιας επιτροπής ε, λαμβάνει υπόψη τόσο σοβαρά την δική μας έκθεση. Είναι πολύ καλή η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα ρουμάνικα για να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Δυστυχώς δεν είχα πολύ χρόνο να εξετάσω πολύ προσεκτικά τα πράγματα. Χτες τα πήρα τα κείμενα ε, και χθες το βράδυ αργά προσπάθησα να δω τι γίνεται με αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες γιατί εμείς είχαμε υποβάλει τις περισσότερες τροπολογίες στην αρχή. Ε, συμφωνούμε με την ομαδοποίηση των τροπολογιών, αλλά όσον αφορά την τροπολογία, τη συμβαστική τροπολογία B, Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να μην συμπεριληφθούν εκεί όλες οι τροπολογίες. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι αποδυναμώνουμε κάπως τα πράγματα με την ε, ε, με την πρόταση αυτή. Παρόλα αυτά μπορούμε να το δεχτούμε διότι ε, επιλύονται πέντε από τα οχτώ προβλήματα τα οποία έπρεπε να επιλύσουμε με ξεχωριστές οχτώ προτάσεις. Παρόλα αυτά θα ήθελα να προτείνω να παραμείνουν κάποιοι όροι εδώ όπως η ένδια διότι στο, στην τροπολογία Δέλτα δεν αναφερόμαστε στη φτώχεια, γιατί δεν καταφέραμε να βρούμε μια συμβαστική λύση, ή στην Ι, ε, όπου εγώ σαν δικηγόρος πίστευα ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε τον όρο ε, ε ο οποίος δηλώνεται στην αστυνομία και να παραμείνουμε στον όρο βιασμός. Ξέρουμε αυτό τι σημαίνει στην εγκληματολογία. Ε, δηλαδή στις, ε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους βιασμούς που έχουν ε, γίνει και στους βιασμούς που έχουν δηλωθεί ή έχουν, για τους οποίους έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση αφετέρου. Τώρα, οι γυναίκες με αναπηρία που δεν μπορούν να μιλήσουν ή δεν μπορούν να ακούσουν έχουν ένα πρόβλημα εκπαίδευσης και παιδεία στη μητρική τους γλώσσα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στη συμβαστική πρόταση D. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και μέσω των τροπολογιών που υποβάλαμε και με τις οποίες, ε, και δεχτήκα, και δεχτήκαμε να ομαδοποιήσουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες ε, πιστεύω ότι καλύπτουμε τα περισσότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες και έστω και αν δεν είμαι 100% ευτυχής με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συζήτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα ο οποίος είναι τόσο σημαντικός. Κυρία Χάρκιν, Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Κώσα για την ε, ε, γνωμοδότησή του. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, μπορούμε να υποστηρίξουμε τις προσθέσεις από τις τροπολογίες. Μία μόνο συμβαστική τροπολογία μας ε, απασχολεί, εκεί όπου επιρρύπτει το βάρος της αποδείξεως στον κατηγορούμενο στο σύστημα του ποινικού δικαίου ε, τουλάχιστον του Ηνωμένου Βασιλείου, το Common Law, αλλά φαντάζομαι ότι θα συμβαίνει το ίδιο και στις άλλες χώρες χωρίς να είμαι ειδική, ε, δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει το, η απόδειξη, το βάρος απόδειξης των κατηγορούμενων. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε τη σχετική τροπολογία. Στο δε σημείο 26. Έχουμε ζητήσει μια προφορική τροπολογία εκεί που γίνεται λόγο για την κατάρτιση για, τους περισσότερους, για τα περισσότερα άτομα με αναπηρίε κατά τρόπον αποτελεσματικό και απλό και ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και εγώ θα ήθελα να βάλουμε τη λέξη ε, ε, ορισμένα κράτη-μέλη, σε αυτό επιμένω, γιατί ζητεί η τροπολογία να γίνεται χωριστά και αποτελεσματικά η κατάρτιση. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει σε σύστημα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα ήθελα σε ορισμένα κράτη-μέλη να προσθεθεί αυτό ο όρο ή σε κάποια κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρο. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Αν όχι, θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Κώσα, θέλετε. Ναι, ευχαριστώ. Δεν, ε, είδα, δεν άκουσα καμία ε, παρατήρηση στην οποία να χρειάζεται να απαντήσω. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία όντω. Ε, σε ό,τι ζήτημα προέκυψε, οι τοποθετήσει των συναδέλφων ήταν πολύ χρήσιμε και με βοήθησαν στη σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών. Όσον αφορά την, ε συμβαστική τροπολογία έγινε μια πρόταση τροπολογίας εχθές που ενισχύει προς την κατεύθυνση αυτή αλλά όντως έχετε δίκιο ότι ε, έχει κάπως ε, αποδυναμωθεί η διατύπωση σε, ως προς ορισμένες έννοιες της τροπολογίας σε άλλα σημεία όμως έχει ε, γίνει πιο αυστηρή. Στη συμβαστική α υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα τα πολλαπλά αυτά μείον εκτήματα και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για τις γυναίκες με αναπηρίες θέλω να υπογραμμίσω ότι το γεγονός ότι είναι γυναίκα και με αναπηρία αποτελεί ένα διπλό επιβαρυντικό παράγοντα. Και έτσι βρίσκεται ε, σε πιο δυσμενή κατάσταση, σε πιο δυσμενή θέση. Για δε τη γλώσσα, τον, ε, την νοηματική γλώσσα, ε, αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματα της κυρίας Κλιμέντη, αλλά εγώ Ω άτομο με προβλήματα ακοής αντιλαμβάνομαι ότι όποιος χρησιμοποιεί την νομιακή γλώσσα πρέπει να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την μητρική του γλώσσα, δηλαδή την νοηματική γλώσσα στην μητρική του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα ήθελα να κάνω και μια πολύ στόμη παρατήρηση. Έχουμε εδώ δύο φίλους από τον Μπενένα σήμερα φοιτητέ στη νοηματική γλώσσα, οι οποίοι στόχο έχουν να γίνουν ε, διερμηνείς της νοηματικής, βρίσκονται εδώ κοντά μας για να παρακολουθήσουν την κατάσταση και να μπορέσουν καλύτερα να ενημερωθούν για την ε, δουλειά μας και να βελτιωθούν στη δική τους δουλειά, στην προσφορά αυτής της υπηρεσίας των ΠΕΝΕΝ, στο άτομα με προβλήματα ακοής. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα, κάνουμε τις θα το συστήσουμε αυτό. Στις 3 Οκτωβρίου θα τοποθετηθεί με την ψηφοφορία η ε, Επιτροπή μας. Τώρα θα παρακαλέσω τον Φιλ Μπένιον να λάβει το λόγο ε, ώστε να μας παρουσιάσει τις συμβιβαστικές του τροπολογίες 10 τον αριθμό. για το σχέδιο νομοδότησης, οικονομία, θέση εργασία και ανάπτυξη μέσω τη περιβαλλοντική πολιτική Έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και εμείς έχουμε την γνωμοδότηση. Έχετε το λόγο κύριε Βέννε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι όντω έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και ιδιαίτερα επικεντρωνόμαστε στην οικοκαινοτομία και τις θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν χάρη σε αυτήν. Ε, θα ήθελα... Είχαμε βρει και πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους και ηγητές νομίζω ότι είναι σαφές ότι καταγράφεται η ε, προσφορά της οικοκαινοτομίας, και δυνατότητα για ανάπτυξη θέσεων εργασία και γενικότερα ανάπτυξη στην περιβαλλοντική από την περιβαλλοντική πολιτική. Ευχαριστώ τους και ηγητές στο σύνολό τους και ελπίζω και οι ψηφοφορίες να επιβεβαιώσουν την πολύ επικοδομητική διαδικασία συνεργασίας και ελπίζω να μας υποστηρίξετε όσο δυνατόν περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ. Κανείς. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή κύριε Σίγητα. Σε λίγο θα ψηφίσουμε και τη δική σας έκθεση. Επομένως, περνάμε τώρα στο σημείο 6 στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση Τσάμπα Σόγκορ για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στη δημογραφία. Πρόκειται για μια ψηφοφορία που θα την υλοποιήσουμε ηλεκτρονικά. και θα μας επιτρέψει να ακυρώσουμε τα αποτελέσματα μιας ευτυχούς διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στη Δημογραφία. Η διαπραγματευτική ομάδα εδώ κατέληξε σε μια καλή συμφωνία. Εμείς λοιπόν θα εγκρίνουμε το κείμενο της συμφωνίας αυτής που επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά του Συμβουλίου στην Κορεπέρ του Σεπτεμβρίου του 2013. Ήταν ανοιχτή ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλη την κάρτα σας. Εγώ έχω μία που δεν δουλεύει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. 37 ψηφίσατε, 38, 37 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία εποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και προχωρούμε, περνάμε στο σημείο 7 σχέδιο γνωμοδότηση ε, της κυρίας Λόπου Φοντανιέ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Πριν την παράγραφο 1 έχουμε μία τροπολογία Μαρίζα Κορνέλισεν. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 4 της Ιδίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, Τζούπερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, Γκουτιέρες Πρέτο, συμβατή, ψηφίζουμε, περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κατόπιν, Παράγραφος 1 για το τροπολογία 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 ζούμπερ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Πάλι παράγραφος 1 συμβεσμός α από 4 ομάδες υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 8. Πέρας. 19 υπέρ, 20 μία ψήφη κατά δεν εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 10, Γκουτιέρες Πρέτο, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 12 ιδίου υπέρ κατά να επαληθεύσουμε για τη 12. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 15 υπέρ, 19 κατά, 6 εποχές, δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 13, Κορνέλισεν, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Πάλι στην παραγραφό 1, τροπολογία 14, κουτιέρες πρέτο, με την προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, ψηφίζουμε όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Συνδεσμός Β. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγωγός 3, συμβασμός C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάλι παραγωγός 3, συμβασμός D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, 24, Γουτιέρης Πυρέτο, υπέρ, κατά, σας απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 3, την παράγραφο 3, τροπολογία συμβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27, η του υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 4, συμβιβασμός F, από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 ζούμπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός G από 4 ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 κορνέλισεν υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Παράγραφος 539. Κορνέλισεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Συμβασμός H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός I. Τρεις ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. J. Από δύο ομάδες. Υπέρ. Κατά αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Ώρας. 25 υπέρ. 15 κατά μια αποχή εγκρίνεται. Η 48 έχει αποσυρθεί. Να ψηφίσουμε πότε το συμβασμό και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με την ίδια παράγραφο, συμβασμός L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν, με την παράγραφο 7, συμβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παραγωγή τροπολογία 59 κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 ζούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 1 στην παρακρο 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν 65 Κορνέλησαν σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα χωρίς τον όρο key, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και ποιος ε, θεωρεί ότι είναι όρος κλειδί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ που είστε που και με βοηθάτε. Λοιπόν, περνάμε στην 66 υπέρ. Κατά αποχές Επαλήθευση. Σφίστε το όλοι, πέρας. Εικοσιμία υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Συνδεσμός ΟΟΥ για την παραγωγή 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην διαπαράγραφο συνασμός πι, από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν 73 τροπολογία της κυρίας Χίρς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 12 να επαληθεύσουμε το 73 μάλιστα. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 26 υπέρ, 13 κατά, δύο εποχές. Έχετε δίκιο. Το 74. Ψηφίζουμε επομένω την τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, επαληθεύσουμε την 81, δεν είναι ξεκάθαρο. Να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 16 υπέρ 19 κατά, 6 εποχέ. Απορρίπτεται. Συμβασμό Q για την παράγραφο 13 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Κατόπιν 85 Κορνέλισεν υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην συγγήτρια. Et euh, Δεν μπορώ παρά να σα καλέσω να εργαστείτε στα πλαίσια τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, ε, έτσι ώστε να υιοθετηθεί αυτή η γνωμοδότηση στο κείμενο που θα προταθεί τελικά στην Ολομέλεια. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο. Και περνάμε στο σημείο 8 για να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση του κ. Κώσα. Γυναίκες με αναπηρία. Παράγραφος 1. Συμβασμός Α από 4 ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια τροπολογία 4 εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέντε χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την περιεκφάνη συμβασμός Β από δύο ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 1, δύο συμβασμούς έπρεπε να ψηφίσουμε. Ξέχασα να σας προτείνω να ψηφίσουμε το συνασμό ΕΦΑ. Από τέσσερις ομάδες έχει προταθεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν, τροπολογία 16, συγγνώμη 13, κορνέλησαν υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε για τη 13. Ψηφίσατε, πέρας. 22 υπέρ, 18 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβασμό C υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός D, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 17, Κοστέλο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό ή e από δύο ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην παραγραφό 5, συμβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά. Κλειβέτη 25 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 25 άρχεται ψηφορία. Ψήφισα το όλοι, πέρας. 17. υπέρ 21 κατά, δύο αποχές δεν εγκρίνεται. Μετά, τροπολογία 26, κλειβέτη, με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28, κλειβέτη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, συμβασμό σε 8 από 4 ομάδες, συγγνώμη 3, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 του εισηγητή με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, ψηφίζουμε την 33 όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 κλειβέτη. Υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Η 35 καταπίπτει, όπως και 36 και 37 και ψηφίζουμε 38 χαούτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου κεντρονικά. 33 pour. 33 υπέρ. Καμία ψήφο κατά τι αποχέ. Συγχαρητήρια κύριε Σίτα. Nous en venons au dernier vote de notre matinée. Να περάσουμε στην τελευταία ψηφοφορία. Σημείο 9. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του κυρίου Μπενιών για την οικοκοινοτομία. απασχόληση, ανάπτυξη μέσα από τις πολιτικές περιβάλλοντος. Μετά την παράγραφο 5, ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία ΑΣ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1. ψηφίσουμε την τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εδώ τώρα θα ψηφίσουμε μια συμβαστική πρόταση που συμπεριλαμβάνει πολλά πράγματα και εκτιμώντας και διάταξη κτλ. Είναι η ε, συμβαστική πρόταση I. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφη 1, η τροπολογία 12, Evelyn Regner, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία συμβιβαστική Α. Την υποβάλλουν τέσσερις ομάδες, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Και μετά την παράγραφο 2 έχουμε στην συμβαστική πρόταση Β, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2 έχουμε τροπολογία 16. Υπέρ Ουγγουρεάνου. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 Σρέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζ. Πριν από την παράγραφο 3 προφανώς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3, συμβαστική πρόταση C, τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, στην τροπολογία 26, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Α, όχι. Για την τροπολογία 26 Σαρή Εσαγιά θα κάνουμε ηλεκτρονική ε, εξακρίβωση. Ψηφίσατε όλοι. πέρες ψηφοφορίας. 18 υπέρ 21 αποχές έχετε απόλυτο δίκιο η τροπολογία 26 δεν εγκρίνεται επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 27 Σρόντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 4 συμβαστική πρόταση D από 4 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στην παράγραφο 5 έχουμε την συμβαστική πρόταση ε, υπέρ. Τέσσερι ομάδε πάλι και εδώ, αποχές ε, εγκρίνεται. Μετά την, τροπολογία, την παράγραφο 5 έχουμε την τροπολογία 35, υπέρ. Κατά αποχές. Λοιπόν, για την τροπολογία 35, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Σαφέστατα. Μετά την παράγραφο 5 έχουμε τη συμβαστική πρόταση F. Ε, 4 ομάδες συζήτησαν υπέρ, κατά, αποχέσεις. εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 5, τροπολογία 38, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, μπαχ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά έχουμε την τροπολο... τη συμβαστική τροπολογία ζ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43, Κίνγκα Κούτσι, υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 44, Κίνγκα Κούτσι, υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Στην, ε, στην τροπολογία 1 της Γιούτα Στάινμπρουκ. Είναι προφορική ε, η τροπολογία, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Μετά έχουμε την τροπολογία 2 του υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και Τροπολογία 3 Κιγκακούτσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 Κιγκακούτσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και εκτιμώντας α η, τροπολογία 5 Γιούτα Στάινμπουργκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την ε, τη λογική έκθεση ε, σκέψη α έχουμε τη συμβαστική πρόταση κα ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη α έχουμε τροπολογία 8 της Elizabeth Schroeder υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ε, πέρασε ψηφοφορία. 38 38 ψήφισαν, 37 υπέρ, ε, κανείς κατά μία αποχή, ε, ε, τον εισηγητή. Όπως η Edith Power έπρεπε να κάνει διάφορα ταχυδακτηλουργικά με την ε, Επιτροπή Δημόσιων Ελευθεριών, πάλι θα κάνουμε μία αλλαγή γιατί θα ασχοληθούμε τώρα με το σημείο 19. Μην φεύγετε. Σημείο 19 και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπουλόν ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης του για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε Κύριε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στην ε, ανάγκη η επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης να περάσει πρώτα από επενδύσεις περισσότερες αλλά και πιο στοχευμένες. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να είναι και διαφοροποιημένες γιατί χρειάζεται η ανάπτυξη και των νέων τεχνολογικών αλλά και η διαφύλαξη της βιομηχανικής κληρονομιάς. Έχουμε μια τεχνογνωσία στην Ευρώπη και εργαλεία που χρειάζονται μια νέα δυναμική για να μας επιτρέψουν να κατακτήσουμε νέες αγορές και να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στη διεθνή σκηνή. Έχω σε ορισμένες ε, τροπολογίες μου επιμείνει στην ιδέα και των ιδίων πόρων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ε, προδιαγραφές για τις προμήθειες, δημόσιες προμήθειες. Έχουμε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες για τις 13 ε, από τις, 16 από τις 43 συνολικά τροπολογίες που έχουμε τεθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα για την εξέβρεση συμβαστικών λύσεων. Υπέστος από τι τροπολογίε των συναδέλφων μου φαίνονται αποδεκτέ, ενδιαφέρουσε. Δύο παρατηρήσει μόνο για δύο τροπολογίε. Η παριθμόν 1, την οποία θα πρότεινα να καταψηφίσουμε, γιατί ήθελα να διαφυλαχθεί το πνεύμα ενό ισχυρού κοινωνικού διαλόγου που ζητεί να καταργηθεί, η λόγω τροπολογία, και 26 η απουσία ε, δικαστικών δεσμεύσεων ως προς την ε, ε, θέση των εργαζομένων. Εδώ υπάρχει μάλλον θέμα μετάφρασης στα γαλλικά γιατί γίνεται λόγος για νομική πράξη και όχι για νομοθετική πράξη. αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία, για, τη βελτίωση που, για τις βελτίωσεις που προσέφεραν στα κείμενα. Ευχαριστώ πολύ Ταρτέν. Δύο λόγια μόνο. Παραμένουν υποσυζήτηση οι συμβαστικέ τροπολογίε. Εκ μέρου τη ομάδα μου είχα την ευκαιρία να διατυπώσω κάποιε παρατηρήσει και επιπλέον αιτήματα προ τον εισηγητή. Κυρίω στην αναφορά στην έκθεση περί αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων του κυρίου Σέρκα. Με χαρά μαθαίνω ότι ο εισηγητής συμφωνεί με πολλές από τις τροπολογίες μας. Έχουμε καταθέσει όντως ούκο και ελπίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία οι συνάδελφοι να τις υποστηρίξουν. Πενιά. Μπένιον. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του στην υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σημαντική μας δείχνει πώς μπορούμε να ε, δώσουμε μια νέα όθηση, να βοηθήσουμε στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας μας, την ανταγωνιστικότητα, την αηφορία στην Ευρώπη. Η εκλογική μου περιφέρεια έχει παραδοσιακή βιομηχανία, βιοτεχνία ε, και γι' αυτό υποστηρίζω οποιαδήποτε μέτρα μπορεί να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων, ε, την επιβίωσή τους και τη διατήρηση των θέσεων και μάλιστα πρέπει να πω ότι βλέπουμε στη δική μου την περιφέρεια μάλλον αύξηση της απασχόλησης το τελευταίο καιρό. Έχω όμως κάποιες επιφυλάξεις ως προς το θέμα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Επιμένω ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να ε, καταστεί υποχρεωτικό μέσα από ένα μόνο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή να γίνει κανόνας ή κανονισμός, γιατί τότε πια πάβει να είναι ε, κοινωνική ευθύνη. Είναι παραδοξολογία δηλαδή το να το επιβάλλουμε μέσω νομοθετήματος. Ωστόσο συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η πρόοδος προς ένα, κοινωνικό, προς ένα σήμα κοινωνικής εταιρική ευθύνης που θα δείχνει ότι είναι ευαισθητοποιημένη μια επιχείρηση. Εγώ μάλιστα είχα την ευκαιρία να συζητήσω και εν και λόγω μάλλον και της ε, κατάρρευσης του κτηρίου των βιοτεχνιών στο Μπαγκλαντές ε, ε, το θέμα αυτό. Αλλά όπως είπατε πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό. Η συμβαστική D μου ικανοποιεί, η B στο μεγαλύτερό της βαθμό, με μια μικρή δηλαδή μόνο τροποποίηση θα μπορούσα να τη δεχθώ γιατί ομιλεί για δικαιώματα που δεν είναι σωστό Επίσης ε, μιλάει για, ε, μιλάει για θέματα που ανήκουν στην ε, επικουρικότητα και άρα θα πρέπει να περιοριστεί αυτή η διεκδικήση περί δικαιωμάτων που δεν εμπίπτουν στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Καλά καλά ούτε στις αρμοδιότητες των κρατών μελών δεν εμπίπτουν. Δεν μπορεί κάποιος που έχει κοπεί σε ένα μάθημα να διεκδικεί το δικαίωμα να επανέλθει στις εξετάσεις και να, να εξετάζεται επαόριστον μέχρι να το περάσει. Είναι παράλογο αυτό. αλλά εν γέννη είναι πάρα πολύ καλή και θετική έκθεση. Γνωμοδότηση. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Qui est Ουδής δεν αρμόδιζε το θέμα αυτό. Ναι, λυπάμαι, αλλά επειδή αντιστρέψατε τα θέματα στην εμέρηση διάταξη, δεν μπόρεσε να προσέλθει ο αρμόδιος για το θέμα αυτό. Ε, καλά, τότε θα ακούσουμε τον κύριο Μπουλόν. Παρακαλώ. Σειρά σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους κυρίους ε, Μπενιόν και Νταντέν, τους δύο φίλοι που πήραν το λόγο σήμερα για την έκθεση αυτή. Δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα το κύριο Τερτέν, άκουσα και τις παρατηρήσεις του κύριου Μπενιών και για πολλές από αυτές συμφωνώ σε ό,τι αφορά την κοινωνική ετικέτα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για τις συμβεστικές τροπολογίες. Δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα να καταλήξουμε σύνδεσμο. Ευχαριστώ. Ja, herzlichen Dank, Philipp. Ähm, in meiner Sprache Ευχαριστώ πολύ, Φιλίπ. Συνεχίζω στη μητρική μου 25 Σεπτεμβρίου έχουμε την εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών. 26 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή. Στην Ήτρε στις 15 Οκτωβρίου γίνεται η ψηφοφορία. Και στην Ολομέλεια συζήτηση και ψηφοφορία στην περίοδο του Νοεμβρίου. Κάτι άλλο. Στο επόμενο θέμα της ημερησής διάταξης. Το υπαριθμών 11. Διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Κυρία Χάρκιν, έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε το βράδυ κάναμε τον τρίτο τριμερή διάλογο και σημειώνουμε πρόοδο. Τέταρτο τριμερής διάλογος ε, θα λάβει η χώρα στις 30 ε, Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε ότι θα είναι και ο τελικός ε, τριμερής διάλογος. Μακάρι να είναι έτσι. Κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα έχουν να κάνουν με τετόριο σε αυτό που λέμε διάφορα μέτρα όπως παίρνουν τους χάρη τα κίνητρα για τους εργοδότες, ε, παραδείγματος χάρη, τα επιδόματα για τους εργαζομένους ε, του EGF, ε, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όταν παρακολουθούν κάποια κατάρτιση, κάποια κρατημέλη. Όπως γνωρίζετε, εξόδευαν έως και 70-80% του συνολικού κονδυλίου από το EGF για τέτοιου είδους μέτρα και υπήρχε μια ισχυρή εντύπωση στο Κοινοβουλίο ότι δεν υπήρχε προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία και ότι έπρεπε να θέσουμε ανώτατο όριο σε αυτές τις δαπάνες. Πρέπει να πούμε ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν χρησιμοποίησαν τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής που Κοσμοποίηση με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάποια κρατημέλη το έκαναν. Ζήτησε το Κοινοβούλιο ανώτατο όριο 25%. Η Κομισιόν ζήτησε 50% και το Συμβούλιο υποστήριξε το 50% όμως ε, δεν καταλήξαμε σε οριστική συμφωνία γι' αυτό, αλλά τώρα έχουμε καταλήξει σε ένα ανατατόριο του 35% και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμφωνία από το Συμβούλιο από αυτού, γιατί το Κοινοβούλιο δεν είναι έτοιμο να πάει πιο πάνω. Πιστεύουμε ότι ήδη έχουμε προχωρήσει περισσότερο από ό,τι σκοπεύαμε. Άλλα σημαντικά θέματα που εκκρεμούν είναι το θέμα των ποσοστών σε χρηματοδότηση. Το Κοινοβούλιο είχε προτείνει τρία διαφορετικά ποσοστά. Καταρχήν για τα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, το Ταμείο Συνοχής, τα κράτη-μέλη που ήταν σε ένα πρόγραμμα ε, και τα κράτη-μέλη ε, ε, θέλανε τα κράτη-μέλη ένα και μόνο ποσοστό συγχρηματοδότησης, αλλά μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε δύο τέτοια ποσοστά συγχρηματοδότησης, ένα γενικό και ένα ακόμη ποσοστό για τις χώρες που συμμετέχουν σε πρόγραμμα και χώρες που εποφελούνται από το Ταμείο Συνοχής. Και εκεί έχουμε περίπου 11-12 κράτη-μέλη. Και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, γιατί υπάρχουν και πολλά ίσουν σημασία, είναι ότι το Συμβούλιο έχει εισαγάγει τους νέους. Αυτό είναι κάτι εντελώ καινούριο και διαφορετικό και δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό κείμενο. Όμως, σύμφωνα με το Συμβούλιο, θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία και έχει εισαγαγεί ένα σύστημα. Αν τα κράτη-μέλη ζητούν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην θα μπορούσαν να κάνουν αίτηση και για ένα μεγάλο αριθμό νέων, δεδομένου ότι αυτοί οι νέοι βρίσκονταν στην ίδια περιφέρεια με τους εργαζομένους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και επίσης αυτή η περιφέρεια θα μπορούσε να υποφεληθεί από αυτά τα κονδύλια το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την πρόταση ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, όμω πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται αυτό με ένα συνεκτικό τρόπο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και του στόχου του κανονισμού. Και προς το παρόν προσπαθούμε να προωθήσουμε μία δέσμη μέτρων, μία πρόταση στο Συμβούλιο που θα επιτρέψει επιτρέψει να υποφεληθούν οι νέοι, μεν, αλλά να σεβόμαστε, όπως είπα, το πεδίο εφαρμογή και τους στόχους. Αυτή είναι η κατάσταση. Προς το παρόν εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλα μικρά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν, αλλά σημειώνουμε πρόοδο και ελπίζουμε ότι θα αρκέσει ένας ακόμη διάλογος, δεδομένου ότι θα συνεργαστεί μαζί μας ε, και το Συμβούλιο γιατί το Κοινοβούλιο από την πλευρά του έχει συνεργαστεί επαρκώς. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θέλει να λάβει το λόγο. Δύο λόγια ακόμα, μια και είμαι σκιώδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα με την πρόοδο των εργασιών και όσα μπορέσαμε να πετύχουμε στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα θέματα τα οποία ήδη συζητήσαμε στα προηγούμενα σημεία, όσα ακούσαμε μέχρι τώρα τέλος πάντων, όσον αφορά τα κεκτημένα ε, ε πιστεύω ότι σε θέματα της ε, αναδιάρθρωσης ε, μπορέσαμε να πείσουμε το Συμβούλιο για το ότι η θέση μας είναι σωστή. Επίσης υπάρχουν κάποια θέματα όπως συγχρηματοδότηση τα οποία και η, βοήθεια για τους νέους. Αυτά είναι θέματα τα οποία, είναι ακόμα, τα οποία συζητούνται ακόμα, συζητώνται ακόμα και πρέπει να τα παρακολουθήσουμε, ιδίως αφορά τη συγχρηματοδότηση για, την, για αυτούς τους διαφοροποιημένους συντελεστές. Δεν είναι κεκτημένο κόμμα, δεν είναι αποφασισμένο, αλλά πρέπει να δώσουμε μια μάχη. Όσον αφορά την ιδιαίτερη βοήθεια για τους νέους, θελήσαμε να υποβάλουμε προτάσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με το Ταμείο ε, για την παγκοσμιοποίηση. Ε, δεν θέλαμε να ε, αλλάξουμε την φύση, αν θέλετε, αυτής της βοήθειας, λαμβάνοντας υπόψη της απολύσεις σε κάποια περιοχή λόγω της κρίσης, λόγω της παγκοσμιοποίησης. Θέλαμε η βοήθεια αυτή να είναι αποκλειστικά για νέους. Αυτές είναι οι απόψεις της ομάδας μας, πάνω στις οποίες θα επανέλθουμε, πιστεύω. Ευχαριστώ Φρέντερικ, κυρία Χάιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Χάρκιν. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, είχατε ε, συζητήσει ε, την πρόσφατη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που ήταν λίγο σκεπτικό όσον αφορά τη χρήση του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση το συζητήσατε καθόλου. Συζητήσατε καθόλου την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Επόμενο, στον κατάλογο των μιλητών είμαι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αναλάβει εσύ τι ε, διαπραγματεύσει, αγαπητή Μάριον. Έχουμε πάσα εμπιστοσύνη στι ικανότητέ σου για τη διαπραγμάτευση ήταν ένα θέμα το οποίο ε, στη Γερμανία ιδιαίτερα δύσκολα μπορέσαμε να πείσουμε τις αρχές ότι είναι χρήσιμο το Ταμείο για την Αντιπαγκοσμιοποίηση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε με όρους συγκεκριμένους και όχι θεωρητικούς γιατί πρόκειται για χρήματα τα οποία ε, πηγαίνουν κατευθείαν στον πολίτη και τον στηρίζουν σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ε, δεν είναι γράμμα κενό, δεν είναι ε, λόγια και υποσχέσεις, αλλά μια πολύ ουσιαστική βοήθεια. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Χάρκιν και της εύχομαι κάθε επιτυχία. Πιστεύω ότι και για τη χώρα σου και για σένα προσωπικά έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο στο θέμα αυτό για να απαντήσω στην ερώτηση της Σάρη. Όντως συζητήσαμε το θέμα της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου και ε, το Συμβούλιο θα το θα λάβει υπόψη κάποιες από τις συστάσεις της έκθεσης. Τρεις συστάσεις ε, έβγαλε το ελεκτικό συνέδριο, αλλά πιο συγκεκριμένη για μας και πιο σημαντική για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, παραδείγματος χάρη. Ε, το, συμβούλ, το ε, ελεκτικό συνέδριο άσκησε κριτική γιατί ε, πιστεύουμε ότι, πιστεύει μάλλον ότι κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν ε, με λάθος τρόπο τα κονδύλια του, των ταμείων. Εμείς ζητήσαμε για τον όριο των 25% ε, και ένα μικρό ποσοστό όμως των κρατών μελών χρησιμοποίησε σημαντικά ποσά των, ταμείων, των διευθυντικών ταμείων για αυτά τα επιλέξιμα μέτρα για δώσει κίνητρα ή και για άλλου είδους μορφή και για άλλης μορφής επιδόματα που δεν ε, προσέφεραν ε, κάποια ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Απλώς ανακύκλωναν τα χρήματα. Γι' αυτό επέμενα σε αυτόν τον όριο των 25%. Το Συμβούλιο και η Κομισιό ήταν ικανοποιημένοι με το 50% και εμείς τελικά αποφασίσαμε ένα μια μέση λύση 35% για αυτά τα μέτρα. Το Συμβούλιο δεν, είχε, δεν μας μπορούσε να εγγυηθεί ότι αυτή θα ήταν η τελική απόφαση, αλλά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων κατέστησα σαφές στο Συμβούλιο και ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό ε, που έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι το Κοινοβούλιο ε, προχώρησε όσο το δυνατόν ε, περισσότερο μπορούσε αυτά. Ευχαριστώ Μάριον, πιστεύω ότι δείχνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αυτό το σημείο 11. Περνάμε στο σημείο 12 τώρα. Η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ganz anderen Platz als sonst. Αλλά κατά θέση μου φαίνεται. I would like to say that um, this item, number 12, θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό, το υπαριθμόν 12, αφορά πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μια οδηγία δηλαδή για την επαναδιατύπωση της οδηγίας του Συμβουλίου ε, που αφορά φοιτητέ και ερευνητές. Στόχος της είναι να προαγάγει κατά το βέλτιστο τρόπο την μεταφορά τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων έτσι ώστε να βοηθήσει και να προσφέρει και εγγυήσει κυρίως σε θέματα ε, δίκαιης μεταχείρισης και κοινωνικής προστασίας σε ομάδες υπηκών τρίτων ε, χωρών. Ήταν ένα δύσκολο θέμα διαπραγμάτευσης. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόταση για τη βελτίωση των διατάξεων που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών, φοιτητέ, φοιτητές, ε, ερευνητέ, εθελοντές, μαθητές, διευρύνεται δηλαδή το πεδίο. Και έχουμε και δύο νέες κατηγορίες υπηκών τρίτων κρατών ε, πρόκειται για άμυστους βοηθούς, ο ΠΕΡ δηλαδή, και έμυστους ασκουμένους, ε, για, για τους οποίους δεν υπάρχει ακόμα νομικά αποδεκτή κοινή ρύθμιση. Αυτό καθιστά πιο περίπλοκο το φάκελο, το θέμα δηλαδή, διότι είναι πιο πολλές οι διαφορές παρά τα κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών των κατηγοριών υπηκών τρίτων κρατών. 80 ντροπολογίες έχουν ε, κατατεθεί από τους χιώδεις εισηγητές, από το ΕΛΚ, τους πράσινους την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ τις εισηγήτριες που έχουν τις συντάκτρες των νομοδοτήσεων οι οποίες εμπλουτίζουν και η κυρία Χίρς και η κυρία Λάμπερτς και η κυρία Σάια με τις τροπολογίες του στα κείμενα. Ε, χτες κάναμε συζήτηση με τις σκιώδεις συγγήτριες σε κάποιους τομείς προτείνω συμβαστικές τροπολογίες και δι. Τρεις αιτιολογικές σκέψεις, 12, 23 και 36, προτείνουμε να ενσωματώσουν συμβαστικές τροπολογίες και αφορούν ε, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο προσδιορισμός των επικών τρίτων χωρών ε, για την αντιμετώπιση τους ως ερευνητών, στις χώρες στις οποίες ε, γίνονται δεκτοί, εγκαθίστανται και στην 23 και 36 έχουμε να κάνουμε με την πρόσφαση φοιτητών στην αγορά εργασίας, όπου ορίζουμε ένα ε, ελάχιστο αριθμό ορών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εργάζονται. Ε, εδώ βλέπουμε αποκλήσεις απόψεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Κάποιες επιμένουν σε 10 ώρες εβδομαδιαίως, άλλες λένε τουλάχιστον 20 και έτσι πρέπει να δώσουμε πιο προσεκτική σκέψη στην υπόθεση αυτή για να καταθέσουμε την προφορική, την συμβαστική τροπολογία. Η τροπολογία υπερθυμών 36 αναφέρεται στην ισότιμη μεταχείριση και την κοινωνική ασφάλιση. Εδώ προσπαθούμε να εξετάσουμε αν, αυτό, αν οι προτάσεις ευθυγραμμίζονται με την οδηγία για την μπλε κάρτα ή ενιαία άδεια παραμονής. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι ισχύει στη σχετικές, ε, σχετική νομοθεσία, μπλε κάρτα, ενιαία άδεια παραμονής και αναλόγως θα προσαρμόσουμε το κείμενο. Έχουμε 13 άρθρα στην ε, πρόταση ε, εδώ. Ε, τα συστήσαμε χθε ε, διεξοδικά. αρκετέ τροπολογίε που αφορούν τα άρθρα έχουν κατευθεί από τις εισηγήτριες που σας ανέφερα και νωρίτερα. Οι 3F, 3I, δηλαδή και 3M, μη έχουν ε, σε ένα αντικείμενο της άμυστες βοηθούς ή τους έμιστους ασκουμένους και χρειάζεται περαιτέρω μελέτη διότι βλέπω μια διαφορετική προσέγγιση από τις πολιτικές ομάδες και με τις κατηγορίες αυτές των υπηκών τρίτων κρατών. Συζητούμε, κάποιες από τις ιδέες μας βρίσκουν σύμφωνους, κάποιες άλλες όχι. Και επίσης εξετάσαμε διεξοδικά άλλα άρθρα, το 6F, σιγματάφ δηλαδή, όπου αναφέρεται πως θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποδέχονται υπηκόους τρίτων κρατών και να τους επιτρέπουν να διαμένουν στην επικράτειά τους με τα στοιχεία που ορίζονται από την πρόταση και που θα παρέχουν οι εργοδότες, όπως είναι αυτοί θέλουν να εργαστούν, συμφωνίες, ε, συμβάσεις ε, και περιεχόμενο τη συμβάσεω εργασία, που ενδεχομένω θα έδινε τη δυνατότητα για παράταση τη παραμονή στη χώρα. Συζητήσαμε το 19α, το 12α, 12β που αφορούν πάλι ειδικέ ε, συνθήκε για του ερευνητέ. και τα ε, δικαιολογητικά που θα χρειάζονταν για να μπορέσει να παρατείνει κάποιο την παραμονή του στη χώρα. Το 14 ειδικέ συνθήκες για τις εσωτερικέ άμεσε βοηθού, χωρί όριο ηλικία. Και έχουμε και κάποια άλλα άρθρα συζητήσει. Ισότιμη μεταχείριση με το άρθρο 21 και 24 ε, για αναζήτηση θέσης εργασίας, διότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική προσέγγιση ως προς την περίοδο παραμονής κατά την οποία δικαιούται να παραμείνει ο υπηκός της ε, χώρας. Υπάρχουν κράτη που λένε ότι μπορούν να παραμένουν για 6 μήνες, άλλα μιλούν για 12 μήνες, άλλα για 18 μήνες που θα επέτρεπαν ταυτόχρονα και την ε, ε, ανάληψη μιας θέσης εργασίας ή την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Έχοντα συζητήσει με, τους με τις χειροδησηγήτριε, θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνία σε κάποια θέματα ή στα περισσότερα είτε με τη μία ε, πολιτική ομάδα είτε και με όλες και επίσης ε, κάποιες ε, τροπολογίες τις οποίες έχω το σημειώσει μη παραδεκτές ή ως αρμοδιότητας Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών δεν μπορώ να κάνω δεκτές. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τη Γραμματεία για την υποστήριξή της. Είχαμε πάρα πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Παρουσία, ε, μας κατατέθηκε αυτή η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις πριν από τις θερινές διακοπές. Η Γραμματεία λοιπόν μας στήριξε σε όλη αυτή την προσπάθεια να προσαρμοστούμε στα πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να προλάβουμε να καταθέσουμε τι ε, προτάσεις Ευχαριστώ τις και όλες και σκοπεύω να καταθέσω τις τροπολογίες, τις συμβαστικές τροπολογίες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή, αγαπητή κυρία Παπαδοπούλου. σα ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ πολύ και για τα ευγενικά σα λόγια προ τη γραμματεία. Είναι κάτι που λησμονούμε συχνά. Ήταν πολύ θετικό το ότι το αναφέρατε. Οι σκιώδει συγκίτριε τώρα, η κυρία Σαλιά εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε χτες για πιθανούς συμβιβασμούς. Είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς γιατί έχουμε ταυτόσιμες απόψεις σε πολλά θέματα. Πολύ καλά έχει θίξει η εισηγήτρια τα θέματα που είναι κάπως επίμαχα και υπάρχουν κάποιες τροπολογίες προς, που πηγαίνουν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ποια γραμμή θα ακολουθήσει η Επιτροπή μας. Όμως, όπως είπε και η συγγήτρια ήδη, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή αυτής της οδηγίας ε, και ε, στους άμεστους ε, ε, βοηθούς αλλά και σε όσους προβαίνουν σε εθελοντική εργασία είτε με αμοιβή είτε χωρίς αμοιβή. Νομίζω ότι είναι κάτι και λόγιο ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτές τις ευάλωτες ομάδες και μπορώ να φανταστώ ποια εκμετάλλευση θα μπορούσε να γίνεται σε σχέση με τις ομάδες αυτές γιατί αν δεν καλύπτονται από μια κανονική σύμβαση εργασίας η θέση τους είναι αδύναμη, πολύ αδύναμη και μάλιστα πολλές από τις δικές μου τροπολογίες ε, στοχεύουν στο να υπερασπίσουν τη θέση αυτών των ομάδων. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να ακολουθήσουμε όσα ακολουθούνται στην ενία άδεια. Έχουμε ήδη ψηφίσει εδώ αυτή την οδηγία. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τα άρθρο 21 και το εκτιμώντας 36. Και το τρίτο ζήτημα είναι ότι κάποιες από τις τροπολογίες μου αφορούν το εξής. Αν υπάρχει αν υπάρχουν ήδη πιο ευνοϊκέ διαδικασίε στα κράτη-μέλη, νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτά τα κράτη-μέλη να τι διατηρήσουν. Όμως, όπως είπε και η συγγήτρια, θα ήταν καλό αν καταλήξουμε σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα στενοχωρό διάγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σκιώδη συγκήτρια εκ μέρου των φιλελευθέρων και αντιπρόεδρο τη επιτροπή μα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τι ευχαριστίες μου προ την εισηγήτρια και τι σκιώδη συγκήτριες από τι άλλε ομάδε. Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα. Λυπούμε που χρειάστηκε να πει έχουμε τόση πίεση χρόνου στην επεξεργασία του, διότι έχουμε να κάνουμε με θέματα που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Τεράστια σημασία για το πόσο θα μείνουν σε ένα χάρο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωση, πόσες ώρες μπορούν να δουλεύουν όλα αυτά. Γι' αυτό είναι πολύ κρίμα που είμαστε υποχρεωμένοι να το επεξεργαστούμε υπό τόση πίεση χρόνου. Επίση, ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου από τρίτα κράτη, οι οποίοι ερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρειάζονται και προστασία από την εκμετάλλευση. Πρέπει να του ε, προστατεύσουμε λοιπόν από την υπερβολική εκμετάλλευση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να του αφήσουμε και ελεύθερου, να αξιοποιήσουν ευκαιρίε που ενδεχομένω του προσφέρονται. Πρέπει λοιπόν, όπω είπα, και την προστασία αλλά και τι ευκαιρίε να του δώσουμε, να μην του στερήσουμε κάποιε ενδεχομένε ευκαιρίε. Ε, αυτό θα είναι η λεπτή ισορροπία στην οποία θα πρέπει να δώσουμε προσοχή. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική γραφειοκρατία ως προς ε, την επιβάρυνση των ερευνητικών ιδρυμάτων στο 12-2 επί παραδείγματι. Για μας είναι περιττό μια επιχείρηση και δεν είναι καν δυνατόν θα έλεγα εγώ ε, μια επιχείρηση, ένα ερευνητικό ίδρυμα να υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Ευρωπαίος πολίτης ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει τα ίδια καθήκοντα κατά τρόπο εξίσου ικανοποιητικό. Δεν νομίζω. Θα μπορούσε να πει ένα ερευνητικό ίδρυμα, μια επιχείρηση. Εγώ ψάχνω τον καλύτερο, αναστώ τον καλύτερο ε, ε, ειδικό, επιστήμονα κτλ. ερευνητή και αυτό να αρκεί. Δεν μπορεί να ζητάμε να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο. Αυτό γραφειοκρατικά θα σήμαινε τεράστια επιβάρυνση και νομίζω ότι μπορούμε με μια πολύ απλή ε, αλλαγή στη διατύπωση να απαλλάξουμε τι επιχειρήσει και τα ερευνητικά ιδρύματα από τεράστιο βάρο. Ένα άλλο σημείο πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι το πόσο μπορούν να εργάζονται οι φοιτητέ. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για 20 ώρες. Οι 20 ώρες είναι πολλές, πιστεύω. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα και πολλές ε, ε, πόλεις και κυρίως πανεπιστημίου πόλεις θα έλεγα, πόλεις με μεγάλα πανεπιστήμια όπως το Λονδίνο, όπως το Μόναχο, όπου είναι τόσο ακριβό το νίκη που χρειάζεται να δουλεύει ο φοιτητή 20 ώρες ή και περισσότερο γιατί διαφορετικά ούτε το νίκη του μπορεί να πληρώσει, πόσο δε μάλλον να εξασφαλίσει την, ε, τροφή του ή ένα βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να μην ε, κατέβουμε πάρα πολύ χαμηλά. Το, οι 33 βέβαια στο 33 μάλλον θα έλεγα ναι τουλάχιστον να αναφέρεται έτσι, αλλά στο 33 παράγραφος 3 και θα ήθελα πολύ προσεκτικά να σας το διαβάσω, λέει ότι κάθε κράτος μέλος ορίζει πόσες ώρες την εβδομάδα ή πόσες ε, ε, ημέρες το χρόνο μπορεί να ασκείται αυτή η ε, δραστηριότητα κατά το μέγιστον και αυτή η δραστηριότητα κατά 20 δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20 ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχο ποσό ε, στο χρόνο. Εάν λοιπόν μιλήσουμε για 10 ώρες εμείς, ουσιαστικά αποστερούμε από πάρα πολλούς φοιτητές τη δυνατότητα της επιβίωσης. Και αυτό είναι για μένα κόκκινη γραμμή. Πρέπει να το συζητήσουμε. Ιδάλλως νομίζω ότι απλώς Μίλαμε για φιλοσικείς δηλαδή τους λέμε ναι ελάτε στην Ευρώπη, αλλά βασικά δεν θα μπορείτε να ζήσετε. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι το πόσο μπορεί να παραμείνει κανείς ε, μετά την περίοδο αυτή. Εμείς τα λέγαμε 18 μήνες, να παρατείνετε δηλαδή παραμονή 18, 18 μήνες, γιατί θέλουμε οι πιο ικανοί, οι πιο ευθύς να μπορούν να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην τους αναγκάζουμε να να φεύγουν, να σου δίνουμε την ευκαιρία να στήσουν ενδεχομένω μια άλλη θέση εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει 12 μήνε μόνο, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα πολύ κακό και αρνητικό μήνυμα για όποιον νέο θέλει να έρθει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η φωνή των φιλελευθέρων, λέει ο Πρόεδρο. Ήταν και πολύ επικριτικά τα λόγια σα. Και τώρα η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της ε, και συμφωνώ με όσους ε, είπαν ε, ότι λυπούνται επειδή πρέπει να εργαστούμε τόσο γρήγορο. Γιατί αν δούμε και το τι συμβαίνει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, εκεί η Επιτροπή είχε προθεσμία μικρότερη για την κατάθεση τροπολογιών και νομίζω ότι και η δική μας Επιτροπή έχει παρόμοια προβλήματα και τελικά μπορεί να καταλήξουμε να μην καλύψουμε θέματα που θέλουμε να καλύψουμε επειδή δεν θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και αυτό είναι πραγματικά τυχές. Επίσης, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν για το ότι δεν πρέπει να πιστοχωρήσουμε σε αυτή την οδηγία. Υπάρχουν δηλαδή κράτη-μέλη που έχουν ε, κάποιες πιο ευνοϊκές διατάξεις, δεν θα πρέπει να τις θίξουμε. Και Έρχομαι τώρα στο θέμα της ισοτιμίας με την άδεια ή με την μπλε κάρτα. Υπάρχουν αυτές οι διαφορές εδώ και έτσι διατρέχουμε τον κίνδυνο να οπισθοχωρήσουμε, να σημειώσουμε επιστοδρόμηση παραδείγματο τόσο σε ό,τι αφορά τα μέλη τη οικογένεια. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμεί ω ομάδα. Και νομίζω τώρα, αν αναζητήσουμε παραλληλισμού με την εννέα άδεια και την κάλυψη εκεί, εγώ επί τη αρχή δεν έχω πρόβλημα για τι πρόσθετε ομάδε, αλλά θα ήθελα να μου πει κάτι κομισιόν, ε, πώ ε, πιστεύει ότι ευθυγραμμίζονται αυτά και αν υπάρχει δεν υπάρχει αποκλεισμό. Κυρίω ε, σε ό,τι αφορά την νέα άδεια, αν καλύπτει όσου εργάζονται και που έχουν το δικαίωμα να εργάζεται και μπορεί κάποιο να πει να καλύπτει και του φοιτητέ αν ε, του δώσουμε το δικαίωμα να εργαστούν. Αλλά <laughs> αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο και βέβαια θα υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν σε αυτό το ζήτημα. Όμως, αν ε, μιλάμε για κάποιες από τις άλλες ομάδες, δεν ε, εξετάζουμε κάτι που κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν σχέση απασχόλησης. Ε, πολλοί θεωρούν ότι ο θελοντισμός δεν είναι σχέση εργασίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα ε, με το ότι εδώ ακολουθούμε την εξή κατεύθυνση. Κάθε κατηγορία αντιμετωπίζεται σαν να πρόκειται να έχουμε παντού σύμβαση εργασίας. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ποια είναι η βάση ε, επί της οποίας έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και αν ε, δραστηριοποιούνται ως οπέρ ή ως εθελοντές και αν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μιλάμε για δίκαιο συμβάσεων και σε κάποιες περιπτώσεις, εκεί όπου γίνεται λόγος για δικαιώματα απασχόλησης είναι σωστό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν εδώ για να μην οθούμε τους ανθρώπους σε μια σχέση απασχόλησης ε, που δεν είναι η σχέση όπως την κατανοούν αυτοί με αυτούς τους οποίους δουλεύουν. Κάποιες ε, από τις τροπολογίες ασχολούνται με ε, τους έμισθους ή άμισθους που, κάνουν πρακτική. Νομίζω ότι για ορισμένα κράτη-μέλη αυτό το θέμα της πρακτικής ε, πολλές φορές θεωρείται ότι είναι συνέχεια της κατάρτισης, μιας εκπαίδευσης. Ενώ για κάποια κράτη-μέλη δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θεωρούν ότι ε, μέσω της πρακτικής οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία πριν να μπουν επίσημα στην αγορά εργασίας. Δεν συνδέεται με τις σπουδέ, δηλαδή. Έτσι λοιπόν η δική μου ομάδα θα είχε προβλήματα να υποστηρίξει τροπολογίες ε, που ουσιαστικά περιορίζουν ε, τους ορισμούς. Το θέμα τώρα για τους ε, τους βοηθούς, για τους ΟΠΕΡ, τέθηκε ένα θέμα ηλικία σε σχέση με το αν έχουμε το άρθρο 3 ή το άρθρο 14. Και πάλι η δική μου ομάδα θα ήθελε να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε υπό ποιες συνθήκες προσλαμβάνονται τα άτομα αυτά. Δηλαδή, αν ε, θέλετε να μην υπερβαίνουμε τα όσα λέει η σύμβαση το αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με το AIDS και με, με την ηλικία, με συγχωρείτε, και με το να υπάρχει ανώτατο όριο για τους όμιστους βοηθούς. Εμείς θα προτιμούσαμε να μην έχουμε ανώτατο όριο. Πιστεύουμε ότι κάποια άτομα μπορεί και αργότερα να θέλουν να βιώσουν ε, αυτή την εμπειρία, να κατανοήσουν άλλους πολιτισμούς. Έτσι λοιπόν δεν θέλαμε ανώτατο όριο ηλικίας εκεί. Όμως ε, εμείς θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες που θα διατηρούν όλα αυτά στο δυνατόν πιο ανοιχτά και ξεκαθαρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων και τις προσδοκίες τους. Όμως ε, θέλουμε να δούμε να επωφελούνται όσο δυνατόν περισσότερα άτομα και να θυμόμαστε ότι εδώ μιλάμε για ένα νομοθέτημα το οποίο θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο για ένα-δύο χρόνια και με αυτό το πνεύμα θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος το λόγο. Όχι. Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις για την πραγματικά ε, πολύ καλή δουλειά που κάνανε για, τις, ε, έκθεση, για την έκθεση και για τις τροπολογίες. Κάποια διευκρινήσεις, κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που έγιναν στην Κομισιόν. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ο στόχος αυτής της, αυτών των προτάσεων είναι κυρίως καταρχάς να μεγαλώσουμε, να αναπτύξουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσελκύσουμε ταλέντα. Τώρα, ε, επίσης, ε, να προωθήσουμε ανταλλαγές ή να προστατεύσουμε άλλες ε, ευαίσθητες ομάδες. Δεν θεωρούμε ότι, είναι, ότι η έκθεση αυτή έχει να κάνει με τη μετανάστευση Κάποιες ομάδες μπορεί να πλήττονται ή να εντάσσονται μάλλον, αλλά δεν μιλάμε εδώ για την εργατική μετανάστευση. Αυτό ξέρω βέβαια ότι εσείς είσαστε Επιτροπή Απασχόλησης και η απασχόληση για σας είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι ομάδες που καλύπτονται από αυτή την έκθεση δεν εμπίπτουν απόλυτα στον ορισμό του labor migration, στη μετανάστευση εργατικού δυναμικού δηλαδή. Αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας όταν εξετάζουμε κάποιες από τις τροπολογίες που μπαίνουν σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες ε, πολλές ε, όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και τον καθορισμό ε, κάποιων στοιχείων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις εργατικές σχέσεις κτλ. Αυτό δεν ήταν, αυτός δεν ήταν ο στόχος της πρότασης της Κομισιόν, να μπούμε δηλαδή σε τόσες λεπτομέρειες όσον αφορά την εναρμόνιση του εργατικού δικαίου των κρατών μελών και αυτό είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο και για το Συμβούλιο για τα κράτη-μέλη. Δεν θέλαμε να μπούμε σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο όμως προτείνουμε, μέχρι σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, όπως κάναμε και σε άλλες προτάσεις για την μετανάστευση, είναι η εναρμόνιση των δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στην ενιαία άδεια και στα δικαιώματα της ε, ισότιμης μεταχείρισης που εμπεριέχονται στην ε, ενιαία άδεια, την, ε, την, την γαλάζια άδεια κτλ. Για να εξηγήσω λίγο λίγο την λογική μας όσον αφορά την ίση μεταχείριση και τη σχέση που έχει με την ε, ενιαία άδεια, γιατί υπήρχαν κάποια ερωτηματικά. Καταρχάς, ε, όσον αφορά τους ερευνητές, ε, βασιζόμενοι στην ισχύουσα οδηγία όσον αφορά τους ερευνητές, οδηγία του 2005, οι ερευνητές δικαιούνται πλήρη ίση μεταχείριση χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς παρεκκλήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία. Και αυτό θεωρήσαμε ότι έπρεπε να παραμείνει. Δεν θέλαμε να υποβαθμιστεί το καθεστώς. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε να παρεκκλίνουμε από το 12β της οδηγίας για την ενιαία άδεια που βάζει κάποια, κάποιους περιορισμούς στην ίση μεταχείριση. Γιατί πιστεύουμε ότι οι, ερευνητές θα πρέπει να διατηρήσουν ε, τα δικαιώματά τους για πλήρη η ισότητα στη μεταχείριση. Όσον αφορά τώρα τους ε, φοιτητές, πιστεύουμε ότι καλύπτονται από την ε, ενιαία άδεια, διότι έτσι όπως ελέγχθη ούτως ή άλλως η ενιαία άδεια καλύπτει και αυτούς που έχουν άδεια εργασίας. Και στην, στην ε, πρότασή μας προτείνουμε οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν και να ασκήσουν και κάποιες ε, ε, εργατικές δραστηριότητες. Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τις ώρες, γιατί δεν είναι ο βασικός στόχος να δουλεύουν, αλλά τέλος πάντων καλύπτονται με την πρόταση για την ενιαία άδεια και θα συνεχίσουν να καλύπτονται με τις παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις που προβλέπει η ενιαία άδεια. Άρα υπάρχει μια αντιμετώπιση που καλύπτεται από την ενιαία. Και μετά έχουμε και τις άλλες κατηγορίες, όπως ε, τους ε, μαθη, τις μαθητείες, τους, εκπαιδευό, τους ε, αυτούς που, ανήκουν σε, που παρακολουθούν μαθήματα, μαθητεία, ε, οι εκπαιδευόμενοι κτλ. Ευτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο να αφορά την πρόσβασή τους στα αγαθά και στις υπηρεσίες με λίγες εξαιρέσεις. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουν βασικά δικαιώματα, τα ίδια δικαιώματα, έστω και αν δεν αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενοι. Αυτή είναι η λογική της πρότασή μας, όπως είπαμε, όπως έχουμε πει και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, είμαστε διατεθειμένοι να ε, διευκρινίσουμε τις, τις ετελογικές σκέψεις ε, έτσι ώστε να ε, ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ποιος καλύπτεται, ποιος δεν καλύπτεται, αλλά αυτή είναι η λογική που στηρίζει την πρότασή μας, όσον αφορά δηλαδή την, ισότη, την ίση μεταχείριση. Μία τελευταία παρατήρηση για τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν για τις πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Προφανώς εμείς έχουμε προβλέψει και το ενδεχόμενο αυτό που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη να ε, υιοθετήσουν πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις, ε, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα. Ε, αν θέλουν να εκχωρήσουν περισσότερα δικαιώματα, τα κράτη-μέλη το έχουν το δικαίωμα αυτό. Όμως είμαστε λίγο προσεκτικοί να το διευρύνουμε σε όλες τις ε, διαδικασίες, ακόμα και τις διαδικασίες ε, υποδοχής, ε, γιατί εκεί θα, κατακαιρματιστούν, θα κατακαιρματιστεί η νομοθεσία, θα μπερδευτούν τα πράγματα. Αυτό θεωρούμε ότι θα είναι εις βάρος ενός σαφούς νομικού πλαισίου που θέλουμε να υπάρχει για αυτές τις ε, περιπτώσεις. Βέβαια τα κράτη-μέλη έχουν ένα κάποιο περιθώριο ελιγμών, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα, επαναλαμβάνω, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να διευρυνθεί η ελευθερία αυτή των κρατών μελών, δηλαδή σε όλα τα άρθρα, διότι θα καταρρεύσει λίγο πολύ το σύστημά μας, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε ένα ε, σύστημα, ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ελκυστικό και σαφές. Θα σταματήσω εδώ επί του παρόντος και αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Σα ευχαριστώ θερμά και για την πληρότητα των συζητήσεων. Τώρα παρακαλώ την Αντιγόνη να μα πει δύο λόγια, αλλά όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα στη μέση διάταξη και 11 θέλουμε να ξεκινήσουμε την ε, ακρόαση. Ευχαριστώ. Uh, Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν ε, τους Κιώδες, ε, γιατί πράγματι είχαμε περιορισμένη περιορισμένο χρόνο και πραγματικά σκεφτόμαστε ότι αυτό το νομοσχέδιο, επειδή θα έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στη ζωή όλων των Ευρωπαίων, πράγματι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Και την επόμενη φορά σε τέτοιου πολύπλοκου φακέλου ζητώ να έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μα ε, γιατί θα θέλαμε να έχουμε περαιτέρω συζητήσει με την Κομισιόν και θέλω να απευθυνθώ στην Κομισιόν και να της πω όσα είπατε τώρα, να μας τα δώσετε γραπτός για τις συγκεκριμένες κατηγορίες το συντομότερο, ως αύριο είναι δυνατόν, για να μπορέσουμε να έχουμε κατά νου ποιες ακριβώς είναι οι διατάξεις της εφιστάμενης και να μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε στις συμβαστικές μας τροπολογίες. Θα ήθελα τώρα να θέσω κάποια σημεία. Ναι. Ε, πράγματι θέλαμε να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες. Αυτή είναι η πρόθεση όλων των πολιτικών ομάδων. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία για να δούμε πώς αυτό στις συγκεκριμένες τομείς κοινωνική ασφάλισης ηλικία και ανάλογα με τη διάρκεια παραμονή στα κράτη-μέλη πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Αλλά α μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσεις ε, στα κράτη-μέλη και το σωστό είναι να μην καταστήσουμε υποχρεωτικές κάποιε από αυτέ τι διατάξει. Ε, γιατί μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτικές πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας και αυτό το τονίζουμε και σε ό,τι αφορά την ανεργία, να πω κάτι. Ναι, η πρόθεσή μας είναι να έχουμε τους καλύτερους υποψηφίους και να βελτιώσουμε ε, τις συνθήκες στην αγορά εργασίας ε, προσλαμβάνοντας τα καλύτερα ταλέντα από τις τρίτες χώρες. Αλλά δεν πρέπει να ε, ξεχνάμε ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα κενά ε, σε ό,τι αφορά την απασχόληση σε κάποιες χώρες όπως Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, ε, Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και οι Ευρωπαίοι προσπαθούν πάρα πολύ σκληρά να βρουν μια θέση εργασία εντό της χώρας του ή να μπορούν να αποφεληθούν τις κινητικότητες, να πάνε στη Γερμανία ή αλλού. Και αν ε, υπάρχουν τόσες πολλές θέσεις ανεργίας πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η καλύτερη ισορροπία Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για τις ανάγκες απασχόλησης, λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω. Θα θέλαμε και την γραπτή απάντηση της Κομισιόν και να μας τονίσει τις διάφορες ε, οδηγίες ε, που υπάρχουν ε, και να αναφερθεί στις συγκεκριμένες διατάξεις και φυσικά θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε συμβασμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δουλέψετε πολύ καλά πιστεύω τις επόμενες ημέρες. 25 Σεπτεμβρίου έχουμε να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Στις 26 του μηνό στην ψηφοφορία η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών ε, ψηφίζει στις 16 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Και τώρα κοιτάω το ρολόι μου. Έχουμε μόνο 6 λεπτά αγαπητή κυρία Μπάουερ για την ε, στρατηγική ένταξη στον Ρωμά. Θεωρείτε ότι μπορούμε να, χειρι... να ανακαλύψουμε το θέμα. Η τα καταφέρνει όλα. Έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστώ όλους όσους ε, στείλατε τις απόψεις σας. Οι περισσότερες από τις ε, τροπολογίες ε, συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικές. Έχουμε δέκα συμβαστικές και προτάθηκαν και συζητήθηκαν χτες. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια ευρύτερη συμφωνία. Φυσικά Ορισμένες ε, είτε είναι εκτός ε, του πεδίου εφαρμογή, είτε δεν μπορώ να τις υφετήσω. Παραδείγματος χάρη ε, την τροπολογία 11 που αφορά τις μετανάστες και όχι τους Ρωμά. Και κάποιες χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις όπως η τροπολογία 13 της κυρίας Κλειβέτη. Δεν την καταλαβαίνω, ίσως να είναι μεταφραστικό το πρόβλημα, όμως δεν κατανοώ εκείνη την τροπολογία. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Ίσως ε, έχω επικεντρωθεί περισσότερο από ό,τι συνηθώ στην απασχολησιμότητα των γυναικών Ρωμά. Και θέλω να ζητήσω από τους ε, αξιότιμους συναδέλφους να διατηρηθεί αυτή η διάκριση μεταξύ της απασχολησιμότητας, της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ε, και των διακρίσεων. Αυτές οι τρεις κατηγορίες αλληλοσυνδέονται μεν, αλλά δεν είναι οι ίδιες δε. Επομένως, ε, στους συμβιβασμούς προσπάθησα να συνδυάσω αυτά τα τρία φαινόμενα, όμως θα ήθελα να ζητήσω να διατηρηθεί αυτή η διάκριση, γιατί το ένα θέμα είναι απασχολησιμότητα, έχοντας περίπτωση χάρη κατά νου ότι έχουμε 32% ποσοστό αναλφαβητισμού στις γυναίκες Ρωμά. Επομένως, ε, ποτέ δεν θα υπάρχουν ε, επαρκείς θέσεις εργασίας ε, για εργαζομένους με χαμηλή εξειδίκευση, χωρίς εξειδίκευση. Και πολλές από τις τροπολογίες, πέρα από τις διακρίσεις, αφορούν και την εκπαίδευση και τον αποκλεισμό. Εγώ είμαι υπέρ των τροπολογιών που αναφέρονται στην ε, πρώιμη εκπαίδευση των παιδιών και που καλύπτουν αυτό το θέμα εκτενώς. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Εργαζόμαστε επί των συμβαστικών τροπολογιών και θα ήθελα να σας ζητήσω ένα feedback ε, μέχρι σήμερα το βράδυ σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Έντιτ, για την γνωμοδότηση. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις σημαντικές πτυχές ε, αυτού του θέματος του φίλου στην ένταξη των Ρωμά. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως να πω για τις τροπολογίες είναι ότι χρησιμοποιούμε μία γλώσσα που δεν δείχνει, δεν αφορά το πρόβλημα για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ε, αντιμετωπίζουν, που έχουν οι γυναίκες Ρωμά. Εάν, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο συστηματική αντιμετώπιση που να εμφανίζεται και στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε διότι η απασχόλησή τους ε, και η, μη απασχόλησή τους τέλος πάντων των, γυναίκων, αυτών ε, έχει να κάνει και με το σχολικό κλίμα, με το γεγονός ότι εγκαταλείπουν νωρί ε, το σχολείο, ότι το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο δεν είναι το καλύτερο, διότι υπάρχει μια δυσπιστία από πλευρά των γονέων και το αποτέλεσμα είναι ότι πολλά, πολλές από αυτά, αυτά τα παιδιά εγκαταλείπουν πολύ νωρίς στο σχολείο. Για να μην μιλήσουμε και για τις, ε, πολύ, τις ε, εγκυμοσύνες που εμφανίζονται πολύ, σε πολύ μικρή ηλικία. Άρα έχουμε ε, πρόβλημα με την γλώσσα περισσότερο και όχι με τις έννοιες. Σήμερα το απόγευμα θα υποβάλουμε κάποιες προτάσεις και βέβαια προφανώς ε, ε, εάν συμβιβαστικές τροπολογίες μας ικανοποιήσουν όσον αφορά την γλώσσα θα τι υποστηρίξουμε. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η συστηματική αντιμετώπιση, αν θέλετε, πιστεύουμε εμείς ε, με αυτή την πιο γενική. Πρέπει να χρησιμοποιείται μια πιο γενική αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Εάν όχι, η Edith Bauer θα ήθελε να απαντήσει. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ε, συνεργαστούμε για να ολοκληρώσουμε τις, τροποποιητικές, ε, τις συμβαστικές τροποποίησεις. Πολύ θετικό πνεύμα επικρατεί. Λοιπόν, θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες στις 25 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου η Επιτροπή Γενικών, ε, Γυναικών. Λοιπόν, τελειώσαμε με, την ημερήσια, με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης που έπρεπε να εξετάσουμε και το επόμενο σημείο τώρα που θα μας απασχολήσει είναι το σημείο 17, όχι, όχι, λάθος, το σημείο 13, 13 η δημόσια ακρόαση που οργανώνουμε με θέμα της, με βάση μάλλον το θέμα της έκθεσης του κυρίου Μάκιντάιρ, είναι εδώ, δεν είναι, ή της κυρίας Μάκιντάιρ, συγγνώμη. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, ξέρουμε πότε θα έρθει, θα περιμένουμε δύο λεπτά για να της δώσουμε την ευκαιρία να έρθει, γιατί δεν μπορεί να γίνει η ακρόαση αυτή την οποία ζήτησε με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, να την ξεκινήσουμε απουσία της. Ζητώ συγγνώμη από όλου, τα μέλη, τους παρατηρητές, τους διερμηνείς, αλλά διαπιστών, θα διακόψουμε για ένα λεπτό μέχρι ότου δούμε που βρίσκεται. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας, διότι και ο Υπουργός ε, και η Συγήτρια. Λοιπόν, στο σημείο 13 ε, έχουμε την ευκαιρία να οργανώσουμε αυτή την δημόσια κρόαση με κίνητρο την έκθεση πρωτοβουλίας υπεύθυνη της οποίας είναι η συνάδελφός μας η κύρια Μάκιντάιρ, για να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία φιλόξενου περιβάλλοντος, ώστε οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι νεοσύστατες εταιρείες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, γενικότερα αλλά και ειδικότερα για την Επιτροπή μας και η μελέτη της έκθεσης της κυρίας Μάκεντάιρ και για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε στο έργο μας ε, θα ακούσουμε τρεις ε, επιφανείς ε, ομιλητές Καταρχάς τον κύριο Μαρκ Χόμπεν, ο οποίος είναι υπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα θέματα απασχόλησης και συντάξεων ο Γιώζεφ Νίμιτς που είναι ε, γνωστός μας ε, γιατί, ε, γιατί είναι πολύ συχνά παρόν στις συνεδριάσεις μας, γενικός ο γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας της ETUC και η κυρία, την κυρία Λιλιάννα Βολονσίσκης που είναι διευθύντρια ε, για τις κοινωνικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την βιοτεχνία. Προτείνω να δώσω το λόγο στους ομιλητές ακριβώς όπως τους παρουσίασα, 10 λεπτά ο καθένας. Πριν όμως θα ήθελα να επιτρέψω στην εισηγήτριά μας να πει λίγα λόγια για το θέμα που, θα, μας απασχολεί το θέμα που θα απασχολήσει την ακρόαση και να εκθέσει και την θέση της Επιτροπής μας μέσα από αυτή την έκθεση, διότι είμαστε εδώ, μην το ξεχνάμε, ε, στην Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων και όχι εσωτερικής αγοράς ή βιομηχανίας. Η κυρία κυρια θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή μας αποφάσισε να οργανώσει αυτή την δημόσια κρόαση και να συντάξει μια έκθεση. Χαίρομαι που έχουμε παρόντες τρεις ειδικού, τρεις εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό και τους ευχαριστώ που ήρθαν. Η ανεργία και κυρίως η ανεργία των νέων είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή Απασχόλησης. Άρα όλοι, ε, όλους μας απασχολεί το θέμα πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα υποστηρίξει την απασχόληση απασχόληση και θα επιτρέψει ε, να δημιουργηθούν, να αναπτυχθεί η οικονομία και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για 20 χρόνια ασχολήθηκα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πριν έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θέλω να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ενδιαφέρουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα ενδιαφέροντα project, παραδείγματος χάρη Think Small First, ε, η πρωτοβουλία αυτή για το σκέψη πρώτα μικρά ε, ή κάποιες άλλες πρωτοβουλίες ε, που έχουν σαν στόχο, παραδείγματο χάρη, να ε, εντοπιστούν οι 10 πιο γραφειοκρατικέ νομοθετικέ ρυθμίσει που επιβαρύνουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θέλουμε να διευκολύνουμε και την ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει επομένω ένα κεκτημένο στο οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε και πάνω στο οποίο να στηριχτούμε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξασφαλίζουν 9 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, Επομένω, υπάρχει και μεγάλο ενδεχόμενο για καινοτομία, για ανάπτυξη και για περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Το 85% όλων των νέων θέσεων απασχόλησης τα τελευταία ε, χρόνια προήλθαν από τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε Μεγάλες προκλήσεις βέβαια που αντιμετωπίζουμε. Π.χ. ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να είναι στην Ευρώπη αυτοαπασχολούμενοι από 40% έχει φτάσει, έχει φτάσει στο 37%. Οι μισοί θεωρούν, φοβούνται ότι μπορεί να χρεοκοπήσουν και πάνω από το 50% λέει ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσει την απαραίτητη ενημέρωση για το πώς θα ξεκινήσει μια τη δουλειά. Βλέπουμε ότι αυξάνεται και ο διεθνής ανταγωνισμός, ο οποίος προωθείται από όλο ένα και πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα, όλα τα επαγγελματικά προσόντα που χρειάζεται ή δεν έχει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Και υπάρχει μια τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ε, θέσεις επασχόλησης ε, εντατική ειδικής, ειδικής εξειδικευμένης απασχόλησης αν θέλετε και ε, πολλές θέσεις ε, μέχρι το 2020 θα χρειάζονται ε, εξειδικευμένες, εξειδικευμένα προσόντα υψηλού επίπεδου και σε γενικότερες γραμμές η, η επιστήμη, η μηχανική, η η μαθηματική δεν πρόκειται να ε, καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας. Βέβαια υπάρχει Υπάρχουν πολλές απόψεις στην Επιτροπή. Άλλοι έρχονται από τις, ε, από τις ε, συνομοσπονδίες, επαγγελματικές συνομοσπονδίες, άλλοι έρχονται από πιο επιπτυγμένες οικονομίες, άλλοι από οικονομίες που έχουν πληγεί από την κρίση, ε, που έχουν μεγάλη ενεργία, άλλοι έρχονται από περιοχές που δεν έχουν μεγάλη ενεργία. Αλλά τέλος πάντων το βασικό είναι πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει το σωστό περιβάλλον και όπου οι εργοδότες θα απασχολούν και ε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτούς που ζητάνε δουλειά. Ε, σαν εισηγήτρια, αυτό το οποίο θα ήθελα για να προετοιμάσω την έκθεσή μου είναι να ακούσω από τους ομιλητές μας πώς ε, η νομοθεσία μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στην απασχόληση. Να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή πώς λειτουργεί η απασχόληση και η εργασία. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κλίμα και τι ε, πρακτικές ή διοικητικές ή κανονιστικές ε, ε, ρυθμίσεις θα μπορούσαν να υιοθετηθούν έτσι ώστε να προωθήσουμε την απασχόληση. Ελπίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι ζωντανή, καρποφόρα και θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες θα μπορέσουμε να ε, συμπεριλάβουμε στην εκθεσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια. Χωρίς να καθυστερήσουμε πλέον καθόλου θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μάρκ Χόμπεν, ο οποίος είναι υπουργό για την απασχόληση στην Βρετανική κυβέρνηση. Το 2012 γίνεται υπουργό και βγαίνετε από το London School of Economics. Λέμε, είναι economy and political sciences όμως, είναι και ε, πολιτικές επιστήμες από οικονομία. Ποτέ δεν το λένε αυτό όμως. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που με καλέσατε να σας μιλήσω σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανεξαρτήτως όμως του από ποια χώρα προερχόμαστε της πολιτικής μας τοποθέτηση. η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εποχή είναι η ανεργία τον Ιούλιο συνολικά η ανεργία ήταν στο 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για, από, για πολλά από τα κράτη-μέλη όμως ήταν πάνω από 20%. Στο Ρωμανό Βασίλειο βλέπουμε μία πτώση στο 7,1% κάτω δηλαδή το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλλά για να ξαναγυρίσουμε στην Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθούμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίε θα δημιουργήσουν θέσει εργασία. Αν κοιτάξουμε από σε ποιου τομεί εμφανίζονται οι, θέσει οι πρόκειται για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ουσιαστικά. Το 85% δηλαδή των νέων θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κατά την προσπάθεια ώστε να ενθαρρύνουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να θεσπιστούν, να αναπτυχθούν, να να μεγεθυνθούν ώστε να δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας, να προσφέρουν σε περισσότερους ανθρώπους θέσεις εργασίας. Κλειδί όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη βεβαίω είναι η εξασφάλιση του καταλλήλου πλαισίου στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο της παρέμβασής μου σήμερα. Θα πω πώς μπορούμε να στηρίξουμε και ε, την θέσπιση των επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα, το κατάλληλο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στη δουλειά που έχει γίνει στο Ρωμανό Βασίλειο που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι τομεί αυτοί. Θα ξεκινήσω όμω από την αγορά εργασία πρώτα. Και υπάρχουν περισσότερε θέσει εργασία λοιπόν από ό,τι στο παρελθόν. Τριάντα περίπου εκατομμύρια άτομα πάνω από 16 χρόνια ηλικία εργάζονται στον Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή έχουμε αύξηση κατά 301.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό σημαίνει για τους ε, τελευταίους μήνες πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας 29.000 σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσει. και από το Μάιο του 2010 έχουμε 1,4 εκατομμύρια νέες εργασίες στον Ηνωμένο Βασίλειο. Τρεις θέσεις εργασίας για κάθε θέση που έκλεινε στον δημόσιο τομέα μετά τα μέτρα λιτότητα που αναγκαστικά εισήχθησαν. Άρα λοιπόν θέση εργασίας στο δημόσιο τομέα δεν μπορεί να δημιουργείται. Πρέπει να αντιμετωπίζονται και τα ε, ελλείμματα των δημοσιονομικών των κρατών μελών. Και άρα αυτό που βλέπουμε στον Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ευελιξία η οποία χαρακτηρίζει την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, η οποία επιτρέπει να καλυφθεί το πρόβλημα της ανεργίας σε σχέση με προηγούμενες ε, κρίσεις που είχαν παρουσιάσει πολύ ψηλότερο πρόβλημα απασχόλησης. η ευέλικτη αγορά εργασία ήταν αυτή η οποία επέτρεψε και τη διατήρηση των θέσεων εργασία και την πρόσληψη ακόμη νέων εργαζομένων με προσωρινέ θέσει εργασία και επέτρεψε τη δυνατότητα για τον άνεργο να δεχθεί την ε, προτινόμενη σύμβαση προσωρινής εργασία, γιατί έβλεπε ότι υπήρχε δυνατότητα να παραμείνει στην ίδια θέση και να μετατραπεί αυτή η σύμβαση σε ε, μόνιμη είδαμε να μετατρέπονται πολλές προσωρινές θέσεις εργασία σε μόνιμες, μόνιμα συμβόλαια. Αυτό δείχνει και την ευελιξία της αγοράς εργασίας. Πόσο σημαντική μπορεί να είναι όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, προσφέρει ευελιξία ένα μαξιλαράκι, ε, ένα δίκτυο ασφαλείας και για την επιχείρηση, η οποία μπορεί να προσλάβει κάποιους εργαζομένους χωρίς να κινδυνεύει να δυσμευθεί σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά ε, σε μόνιμες θέσεις εργασία, ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει ε, τις προσωρινές αυτές τις εργασίες να τις μετατρέψουμε σε μόνιμες όταν τα πράγματα πάνε καλύτερα για την οικονομία και την επιχείρηση. Στο δανεισμό τώρα. Η οικονομική κρίση είχε σε συνέπεια για τις τράπεζες να διστάζουν να δίνουν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό εισήχθη ένα σύστημα χρηματοδότησης για την ε, προσφορά δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή μειώνουμε το κόστος για την τράπεζα στην ε, παροχή δανείου και αντίστοιχα και στο επιτόκιο, επιδοτείται το επιτόκιο για την επιχείρηση. Προσπαθούμε επίση να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να πούμε ότι ο επιχειρηματίας θεσπίζει μια νέα επιχείρηση και αλλάζει πολλά πράγματα είναι ακριβώ η βοήθεια στην επιχειρηματικότητα, η στήριξη στην υλοποίηση μια νέα ιδέα και στη χρηματοδότηση και τη στήριξη όταν αυτή η επιχείρηση έχει ήδη θεσπιστεί και λειτουργεί. 2.000 επιχειρήσει λοιπόν που δημιουργούνται κάθε μήνα στο ΗΠΑ Βασίλειο που, ε, θεσπίζονται, που ιδρύονται από πρώην ανέργους που να σας ξέρω ένα παράδειγμα τη Χέιλι από την ε, Δυτική Ουαλία που γνώρισα τον προηγούμενο μήνα, η οποία ήταν άνεργη και η οποία άνοιξε έναν βρεφονιπιακό σταθμό που ονομαζόταν Alliance Den, ε, ονομάζεται Alliance Den και μπόρεσε μέσα σε αυτό το πολύ σύντομο διάστημα από την ώρα που άνοιξε το βρεφονιπιακό σταθμό να να προσλάβει και άλλες ε, πάνω από 20 εργαζόμενες, οι οποίες ήταν, ήταν όλες άνεργες. Εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δημιουργούνται έως και 26.000 τελευταίο χρόνο. Ε, έχουμε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που προσφέρει η κυβέρνηση που μειώνει την, ε, το κόστος για τη θέσπιση μιας νέας επιχείρησης που επιτρέπει την λειτουργία χωρίς επιβαρύνση γραφειοκρατική ε, για τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα είχαμε ένα κανόνα ε, μία συν, μία πλην. Με την έννοια ότι αν ένας κανόνας επέβαλε επιπλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, ε, τότε αντίστοιχα εισαγόταν άλλο νομοθέτημα το οποίο μείωνε σε άλλο τομέα την γραφειοκρατία στον ίδιο βαθμό αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιορίζεται η γραφειοκρατία γιατί αυτό σημαίνει ε, πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που μπορεί να χαθούν μόνο και μόνο επειδή υπάρχει γραφειοκρατική επιβάρυνση. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εάν ε, αξιοποιούνταν ο κανόνας one in one out, δηλαδή ένας, ένα, ένας νόμος που επιβαρύνει και ένας νόμος που ελαφρύνει γραφειοκρατικά την ε, θέσπιση και λειτουργία επιχειρήσεων. Επίσης, εμείς τρεφήκαμε και προς επιχειρήσεις, ε, επιχειρηματίες για να τους ρωτήσουμε τη γνώμη τους, να ρωτήσουμε πού βλέπουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και πώς θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε, τις επιχειρήσεις, ώστε να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση, η κανονιστική, η ρυθμιστική, ώστε να στηριχθούν η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη. Αυτή η μεγάλη πρόκληση επέτρεψε στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν τουλάχιστον 250.000 ε, ευρώ το χρόνο και έτσι να αναπτυχθούν και να προσλάβουν πιστούς εργαζομένους. Μια ανεξάρτητη πολιτική, ρυθμιστική, επιτροπή ρυθμιστικής πολιτικής επίσης θεσπίστηκε και παρακολουθεί την, ε, τις συνέπειες ε, της εισαγωγής της νέας νομοθεσίας. Χρειάζεται μια πολύ αυστηρή διαδικασία ε, Παρακολούθηση των εξελίξεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει κάθε νομοθέτημα στην ε, γραφειοκρατική επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να βγάζουμε ιδέες από το μυαλό μας έτσι. Και έτσι αναλόγω γίνονται προτάσει και προ τα Υπουργεία για την αλλαγή τη νομοθεσία. Πρέπει να σα πω όμω ότι ε, τα όσα γίνονται σε επίπεδο μια χώρα μέλου δεν σημαίνει ότι έρχονται σε αντιπαράθεση με τα όσα γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ότι είναι αντίθετα με αυτά. Υπάρχουν πολύ καλέ ιδέε και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και για την υγεία και ασφάλεια. Ξέρετε ότι έχουμε ιδιαίτερο θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο με μια πολύ αυστηρή διαδικασία ε, που εισαγάγαμε για να περιορίσουμε τη γραφειοκρατική επιβάρυνση χωρίς όμως να υποβαθμιστεί η προστασία του εργαζομένου. Και κάνουμε τη διαδικασία της προσαρμογής στους κανόνες πολύ πιο απλή και διαφανή, αλλά ταυτόχρονα δεν ε, είναι λιγότερο ασφαλή δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιθέτως είναι ένας από τους πιο ασφαλείς χώρους εργασίας. Υπάρχει επίσης μια πρόταση για περιορισμό του, της κανονιστικής οικονομικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, πρόταση την οποία θα δούμε και πριν από θα, θα διευκρινίσουμε πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τρόπους να ενισχύσουμε την ε, διαδικασία για καταχώρηση, κατάθεση της αιτήσεως για τη θέση μιας επιχειρήσεως, αλλά πάλι με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία που σας μίλησα, για την οποία σας μίλησα στη Δυτική Ουαλία ε, έχει 17 υπαλλήλους. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να ε, λειτουργήσει η νομοθεσία σε τόσο μικρές επιχειρήσεις. Γιατί αυτή, κυρία, όσο μεγαλώνει η επιχείρηση, τόσο πιο πολλές δυσκολίες θα έχει και τόσο πιο πολύ μεγάλο νομοθετικό πλαίσιο ε, στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί. Η διατήρηση λοιπόν και τα εργασία παραμένει ευθύνη των επιχειρήσεων, όπω είπαμε, όπω ήταν και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Εμεί όμω ω νομοθετική αρχή, ω ε, εκτελεστική εξουσία, έχουμε καθήκον να ενθαρρύνουμε την ε, δημιουργία νέων επιχειρήσεων και να μην την, να μην την ε, καταστήσουμε πολύ δυσκολότερη επιβάλλοντας νομοθετήματα πολύ δύσκολα. Μην ξεχνάμε τις δεκάδες χιλιάδες των νέων ενέργων στην Ευρώπη που δεν μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας Έχουμε καθήκον προς αυτούς να αναλογιστούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και το κόστος της δημιουργίας της ενοργασίας, της σύστασης επιχειρήσεων και τις προοπτικές για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε και για τις προτάσεις που υποβάλλατε. Θα δώσω τώρα το λόγο για 10 λεπτά στον κύριο Γιώσεφ Νίμικ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως ε, αν δούμε τα πράγματα από την ευρωπαϊκή σκοπιά θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη την ε, ποικιλομορφία των καταστάσεων, ε, δηλαδή η θετική περιγραφή του τι συμβαίνει σε μια χώρα θα πρέπει να ειδωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και δυστυχώς εμείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν είμαστε αισιόδοξοι γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ουσιαστικά αποδομούνται οι θέσεις εργασίας, καταστρέφεται η απασχόληση. και με τον ε, ίδιο τρόπο βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα για την οικονομική ανάπτυξη. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μια στρατηγική, την Ευρώπη 2020, για την ανάπτυξη, για την οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είδαμε όμως ε, πώς αυτή η φιλοδοξία να μπορέσουμε να δούμε δημιουργία θέσεων εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υλοποιήθηκε. Όμω ε, το αντίθετο έχει γίνει, η καταστροφή τη απασχόληση. Έτσι λοιπόν, εμείς λαμβάνουμε υπόψη τις εμπειρίες ε, των τελευταίων ετών και διαπιστώσαμε ότι η κρίση αλλά κυρίως η απάντηση της Ευρώπης ε, στην κρίση τελικά δεν εξυπηρετούν μακροπρόθεσμους στόχους. και την κατάσταση αυτή θα πρέπει να τη δούμε με ένα διαφανέ πνεύμα, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικέ εμπειρίες που μπορεί να λαμβάνουν χώρα σε κάποια κράτη. Αν δούμε τα πράγματα από αυτή την οπτική, και μιλώ ως ένας κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί τους εργαζομένους, νομίζω ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να επανερχόμαστε σε όσα είπαμε μαζί με τους εργοδότες όταν κάναμε την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας το 2007 πριν από την κρίση. Εκεί υπήρχε μια προσέγγιση που μας επέτρεπε να προσεγγίσουμε τα ουσιαστικά θέματα για την απασχόληση στην Ευρώπη αλλά και για την ανάπτυξη και το περιβάλλον των επιχειρήσεων με έναν τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πτυχές και φυσικά προσθέτουμε και την δυνατότητα σύγκρισης των εθνικών καταστάσεων. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί εκ νέου πρέπει να ξαναδούμε τις μελέτες αυτές, τις αναλύσεις αυτές και να εξαγαγούμε για κάποια διδάγματα. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό για μας είναι να αναγνωρίσουμε ότι στην προσέγγιση αυτή και κυρίως στις συστάσεις λέγεται ότι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ευνοϊκή κατάσταση στην Ευρώπη έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού έχοντας ως ε, αντιπαλωτέως τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ανατολική Ασία εμείς ε, δώσαμε έμφαση, θέσαμε ως προτεραιότητα την επένδυση στα άτομα. Επίσης, έχουμε εστιάσει σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ασχοληθήκαμε όχι μόνο με τα θέματα της ε, ενεργούς πολιτικής της αγοράς εργασίας αλλά και με τα μακροοικονομικά ζητήματα και εκεί επιμείναμε στην αναγκαιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθούν αντικυκλικές πολιτικές υπογραμμίσαμε και τη σημασία του να επενδύει κανείς στις δημοσίες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος κοινή ωφέλεια. Κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και κάτι που ήταν πρωταρχικό για μας, επιμείναμε στο εξή. Σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που πρέπει να ευνοεί την δημιουργία επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιοτικών, να δημιουργήσουμε έναν ανταγωνισμό σε ισότιμο επίπεδο με ίδιους κανόνες. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα τη αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Ομοθεσία. Φυσικά και εμεί συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα, όμως το ουσιαστικό είναι να μην ε, μειώσουμε την προστασία των εργαζομένων και σε μια κατάσταση κινητικότητας ε, να εξασφαλίσουμε ότι όσοι εργαζόμενοι μεταβαίνουν σε άλλες χώρες την χάνουν ίδιας μεταχείρισης. Έτσι λοιπόν σε όλα αυτά πρέπει να βρούμε την ορθή απάντηση και σε τέτοια είδη μεταρρυθμίσεων όταν ε, μιλάμε για ε, τη λειτουργία των επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη, θα πρέπει και οι κοινωνικοί εταίροι να καθορίζουν, να διαμορφώνουν αυτή την νομοθεσία. Νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον και των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων. Αυτό είναι το ουσιαστικό στο μήνυμα που θέλουμε να διαβιβάσουμε. Και αν δούμε την εφαρμογή αυτών των συστάσεων στα πλαίσια της συμφωνίας που συνάψαμε με τους ε, εργοδότες, αν δούμε τι συνέβη, διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρχε ούτε υπάρχει αυτή η ισορροπία στις ευρωπαϊκές ε, πολιτικές σήμερα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και είναι πάρα πολύ ενισχυτικό γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών και ιδίω των εργαζομένων στο μέλλον του ευρωπαϊκού Οικοδομήματο, αλλά και κυρίω στο δικό τους μέλλον, στην ε, θέση εργασία τους, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, το πρωταρχικό ζήτημα. Και γι' αυτό εμείς ε, δώσαμε μια διαφορετική απάντηση για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, προτείνοντας μια κοινωνική σύμβαση, ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα έγγραφο που νομίζω έχει διανεμηθεί και εδώ, νομίζω ότι το έχετε δει, σας έχει γνωστοποιηθεί. Θα ήθελα να επανέλθω στη συνέχεια σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα που ήταν στην ανάλυση της αγοράς εργασίας και που αναφέρονται και σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο. Ας δούμε καταρχήν κάποιε πολύ σημαντικέ αλλά απλέ ερωτήσει. Κύριε Υπουργέ, εσεί αναφερθήκατε στο πόσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία. Είναι μια μεγάλη ανησυχία αυτή και για τι επιχειρήσει, το γνωρίζουμε. Δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι η συνάδελφο που εκπροσωπεί τι μισέ και μισέ επιχειρήσει που θίγονται περισσότερο θα μιλήσει για το θέμα αυτό, αλλά και εμεί ανησυχούμε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και στα πλαίσια της κρίσης που είναι σε θέση να παράγουν και να προσλαμβάνουν άτομα αλλά δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και υπάρχει ανισότητα στην επικράτεια την ευρωπαϊκή. Παραδείγματο χάρη στη Γερμανία έχουν πρόσβαση επιχειρήσει στη χρηματοδότηση ενώ σε άλλε χώρε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται λοιπόν ευρωπαϊκή δράση για να δοθεί απάντηση. Δεν αρκεί να αναλαμβάνεται δράση σε κάθε κράτο μέλο γιατί κάποια κράτη δεν έχουν τα μέσα. Και αυτή είναι η πρότασή μα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Συμβόλαιο την Ευρώπη, γιατί εκεί αναφερόμαστε σε απαντήσεις που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένουμε στην αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης του τραπεζικού συστήματος για να δοθούν κάποιες απαντήσεις, αλλά και στην καλύτερη χρήση των υφιστάμενων μέσων, το χάρη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματική σε αυτά που κάνει και να έχει περισσότερα μέσα. Ήθελα λοιπόν να αναφερθώ και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο των μεμονωμένων κρατών μελών. επέμενα στο θέμα των ικανοτήτων και των προσόντων. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι για το θέμα αυτό, είναι ζωτικό. Το είπαμε και στην ανάλυση της αγοράς εργασίας και το επεγράμμισε και ο κύριος Υπουργός, αλλά ας δούμε τι συμβαίνει σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις ε, που δεν καλύπτονται. Αν όμως θέσουμε την ερώτηση στα μέλη μας, μας λένε «Μα ο μισθός που προσφέρεται δεν ανταποκρίνεται όχι μόνο στις προσδοκίες, αλλά και στη δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες ενός ατόμου και της οικογένειάς του». Έτσι λοιπόν το θέμα του ύψους των μισθών σε σχέση με τις οι ικανότητες και τα προσόντα του εργαζομένου είναι ένα ζήτημα. Αλλά το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχεται πάρα πολλούς Ευρωπαίους, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη. Το ξέρω γιατί και εγώ ως Πολωνός έχω μια σχετική εμπειρία βάσει των επαφών που έχω στην ε, χώρα μου, στην πατρίδα μου. Όμως εμείς δεν χρησιμοποιούμε πάντοτε με το πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δεξιότητες και τα προσόντα των ε, ατόμων. Πολλές φορές ε, ε, δεν προσφέρουμε την κατάλληλη θέση εργασίας σε ανθρώπους που έχουν πολλά προσόντα και επομένω, πραγματικά πρόκειται για μια τεράστια σπατάλη αυτής της επένδυσης που έχουμε κάνει στα άτομα. Έτσι λοιπόν ας δούμε αυτό το θέμα της μεταχείρισης των ανθρώπων και της εκούσιας ε, κινητικότητας και να δούμε και το θέμα του value for money. Έχουμε επιμείνει σε αυτό, αλλά έχουμε επιμείνει και στο πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις σε αυτές ε, τις ε, δεξιότητες. Γιατί εμείς δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μείωση σε αυτόν τον τομέα. Και τελικά όλα πέφτουν πάνω στους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε απαντήσεις και εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις, πώς θα τις χρηματοδοτήσουμε. Γι' αυτό θέλουμε να συμπληρώσουμε αυτές τις προτάσεις του Κοινωνικού Συμβουλίου και με πιο πιο συγκεκριμένη πρόταση για ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αλλά και για να γίνουν επενδύσεις στους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω πολύ σύντομα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε πιο συγκεκριμένες ιδέες, δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να βρούμε τα κατάλληλα κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο μαζί με την ιδέα ότι δεν πλέπει... Ε, να βλέπουμε τις χώρες που έχουν πετύχει μόνο, αλλά πρέπει να θέσουμε στο στόχο και τις χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω της κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην τελευταία προσκεκλημένη μας, την κυρία Βολοζίνσκη, η οποία εκπροσωπεί την Ένωση Βιοτεχνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είπε και ο Υπουργός, είναι μία από τις βασικές ε, ε, προκλήσεις της ε, Ευρώπης που είναι η έλλειψη ανάπτυξης και έλλειψη απασχόλησης και οι συνέπειες που έχουν στην κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση στην Υπηρό μας γιατί υπάρχουν και βασικές διαφορές και στα κράτη-μέλη. Ο βασικός τίτλος της ακρόασης είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ένα ε, έφορο αν θέλετε περιβάλλον έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, όχι μόνο οι μικρομεσαίες. Και όπως είπε και η συγγήτρια, εφόσον οι μικρομεσαίες είναι ο βασικός, η βασική πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τεθούν στην καρδιά της νομοθεσίας για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία που αφορούν την, ε, ε, την, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 23 εκατομμύρια απασχολεί ε, ε, επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 99,8% μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 18 εκατομμύρια απασχολούν λιγότερο από 10 άτομα. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκπροσωπούν το 60% της προστιθέμενης αξίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, έχουν δημιουργήσει την τελευταία δεκαετία το 85% των νέων θέσεων απασχόλησης και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι 50% από τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιχειρήσεις ενός ατόμου, είναι αυτοαπασχολούμενοι δηλαδή παρά την κρίση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ακόμα η πλέον δυναμική δύναμη ε, για την, ε, στις οικονομίες μας για την ε, δημιουργία απασχόλησης. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να βγει από την κρίση και για να γίνει αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν οι ακόλουθες δράσεις. Η πρώτη είναι να δημιουργηθούν κανόνες. Το να δημιουργήσουμε κανόνες σημαίνει κατάλληλες μακροοικονομικές πολιτικές για να προστατεύσουμε τις ε, επενδύσεις. Όταν μιλάμε για μακροοικονομικές, δηλαδή πρέπει να έχουμε στέρεες φορολογικές πολιτικές και ανάγκη να ε, είναι στέρε και, και υγιής η οικονομία των κρατών μελών και θα πρέπει να μειωθεί το χρέος των κρατών μελών και των ε, ε, οικογενειών. Ε, δεύτερον, είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει ε, πρόσβαση σε επιστώσεις ε, όπως προβλέπονται από το, πρόγραμμα τα και ορίζοντας 2020. Επίσης ε, θα πρέπει να προωθήσουμε την ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τομέα της καινοτομίας. άλλα μέτρα αφορούν την πρόσβαση στις αγορές θα πρέπει να βελτιώσουμε την δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στην αγορά, όχι μονάχα την τοπική αλλά και την διεθνή αγορά. Τέταρτο στοιχείο, για να δημιουργήσουμε αυτό το φιλικό περιβάλλον, είναι η υποστήριξη μάλλον ε, διαθεσιμότητα υπηρεσιών υποστήριξης και ε, αποτελεσματικοί ενδιάμεσοι οργανισμοί. Και όχι μονάχα για τις ε, παραδοσιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τις startups επιχειρήσεις. Πρέπει να έχουν ενδιάμεσες ε, ε, υπηρεσίες υποστήριξης. Η δημιουργία όμως θέσεων επασχόλησης δεν θα γίνει εάν δεν υπάρξει και μια υποστήριξη είναι επιχειρηματικότητα και θα ήθελα να υπάρξουν επομένως νέες συμφωνίες ανάμεσα στους ε, Ευρωπαίους εταίρους. <clears throat> Θα πρέπει να εντοπίσουμε την επιχειρηματικότητα σαν, μία από τις τέσσερις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρχουν και το επιχειρηματικό πνεύμα θα πρέπει να αναπτυχθεί ήδη από τα σχολεία. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει και ένα κανονιστικό περιβάλλον το οποίο να υποστηρίζει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το είπε και η συγγήτρια, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν από άχρηστη, από περιττή γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να εφαρμόσουμε και να σεβαστούμε την πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συζητάτε σήμερα στην Βιέννη για την, για την, σχετικά με την αναθεώρηση και πρέπει να έχουμε μία συνεπή εφαρμογή της αρχής Think Small First που ακόμα δεν εφαρμόζεται βέβαια και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο και το σημείο αφετηρίες για όλες ε, τις ε, νομοθεσίες, καινούριε ή, ή μεταρρυθμιστικές νομοθεσίες πρέπει να είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αντί να ε, υιοθετούμε εξαιρέσεις για αυτές τις νομοθεσίες θα πρέπει αντίθετα όλες οι νομοθεσίες να ε, συμπληρώνονται με ένα τεστ αν θέλετε για την εφαρμογή τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει όλα αυτά, όλες αυτές οι αρχές να χρησιμοποιούν, να εφαρμόζονται μάλλον ε, με συνέπεια. Η εφαρμογή των αρχών αυτών θα περιορίσει την ανάγκη για εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα περιορίσει σημαντικά το διοικητικό άχθος. Λοιπόν, αυτά αφορούσαν το γενικό πλαίσιο. Τώρα θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για τις ε, θέσεις απασχόλησης που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να, να... μπορούν να προσλάβουν κόσμο εάν να το επιτρέπει η αγορά, εάν να μπορούν να στηριχθούν σε εξειδικευμένη εργατική δύναμη. Εάν η αγορά εργασίας είναι αρκετά ευέλικτη και εάν οι μισθοί ε, ευθυγραμμίζονται με την παραγωγικότητα, εάν και εφόσον ο οι φόροι και τα επιδόματα ε, δεν ε, επιβάλλουν κυρώσεις στην, στις επιχειρήσεις, τότε οι θέσεις απασχόλησης θα προωθηθούν, θα αυξηθούν. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τις μικροεπιχειρήσεις, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρχάς να υποστηρίξουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουμε την λειτουργία των αγορών εργασίας και την ανταγωνιστικότητα μέσω του συντονισμού των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει μια καλή διακυβέρνηση από πλευράς των κρατών μελών και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουμε μέσα στα πλαίσια της μικροδιακυβέρνησης και της κατευθυντήριας γραμμές για τη λειτουργία των κοινωνικών εταίρων. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει η σωστή οικονομική υποστήριξη, καταρχάς για ε, επένδυση στην, ε, στην εκπαίδευση, ε, επιδότηση της εκπαίδευσης, υποστήριξη της εκπαίδευσης, όλες, ε, όλων των μορφών, ε, όλες τις μορφές μαθητείας, ε, προσαρμογή στην αλλαγή, η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μπορούν να, να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται αν θέλετε, να μπορούν να προσφέρουν συναχή εκπαίδευση και κατάρτιση. Επίσης, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας που υπάρχει ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στα πλαίσια του προγράμματος EEAPMAE e e, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα τα οποία ψάχνουν δουλειά, να μπορούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση, να τους υποστηρίξουμε οικονομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε. Ένα άλλο θέμα είναι η κινητικότητα των εργαζομένων. Όταν μιλάμε για την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να προσαρμοστούν οι ανάγκες της αγοράς και των εργαζομένων, προσαρμόζοντας τα προσόντα στις ανάγκες της αγοράς και μπορούμε να ζητήσουμε να χρησιμοποιείται καλύτερα το EURES και τα κράτη-μέλη να, είναι πιο, να εφαρμόζουν αρχές διαφάνειας όσον αφορά τις ε, κενές θέσεις που υπάρχουν. Εν κατακλείδη επίσης ε, υπάρχει και η αρχή Think Small First. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα, κυρίως όσον αφορά την νομοθεσία οι προσπάθειες οι οποίες έχουν ε, καταβληθεί από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο μείωση 25% του διοικητικού άχθους πιστεύουμε ότι θα πρέπει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η, η απλούστευση θα πρέπει να είναι σημαντική. Δεν μπορούμε απλώς και μόνο να αναφέρουμε νούμερα χωρίς να περάσουμε και σε πράξεις. Επίσης το κεκτημένο θα πρέπει να υποφεληθούμε από το κεκτημένο και να δούμε κατά πόσον τα νομοθετικά κείμενα που ήδη έχουν υιοθετηθεί, μήπως δημιουργούν προβλήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια που ε, ελπίζουμε ότι μέσα στην, στα πλαίσια της νέας στρατηγικής θα απλουστευθούν περισσότερο και θα εστιαστούν περισσότερο στην πρόληψη και στην καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αντί να προσθέτουν νέους κανονισμούς. Επίσης, το χρόνο εργασίας χρειάζεται να επιλύσουμε το θέμα ε, της παρουσίαση απασχόλησης, ε, του χρόνου απασχόλησης των ε, εργαζομένων. Επίσης, θα πρέπει να ε, ρυθμίσουμε το θέμα της ευελιξίας και της περίοδου αναφοράς. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας για την μετακίνηση των εργαζομένων, την απόσπαση των εργαζομένων, ε, μας ε, απασχολεί κυρίως η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άνθρωπο 12 να δημιουργηθεί μια ενιαία κοινή ευθύνη σε, σε όλα τα ευρωπαϊκά επίπεδα για όλους τους τομείς. Αυτό Μήπως μπορείτε να ολοκληρώσετε. Τρεις γραμμές έχω να πω ακόμα για την ε, απόσπαση των εργαζομένων είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό το οποίο, ζητήσουμε, το οποίο ζητάμε και χρειαζόμαστε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Και ζητώ συγγνώμη που σας διάκοψα και σας πίεσα, αλλά το ρολόι μας ε, πήρε με μια κάποια καθυστέρηση. Ας δούμε λοιπόν τους ομιλητές. Η εισηγήτρια φαντάζομαι θα στείλει το λόγο τελευταίο. Κύριε Ανδρέας Παρέα, παρακαλώ τότε να λάβει το λόγο. Είναι η συγγήτρια από την Επιτροπή Βιομηχανίας, η οποία συμμετέχει ως συνδεδεμένη επιτροπή μαζί με τη δική μας διαδικασία για την έκθεση πρωτοβουλίας. Και στη συνέχεια, κύριε Πλευδιάσικα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η εισηγήτρια σε συνεπόφαση με την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ όσους ε, πήραν το λόγο τους προσκεκλημένους μας σε αυτήν την Επιτροπή, καθώς ε, και το έργο της εισηγήτριας. Και θα είμαστε σε επαφή σε λίγο. Εδώ έγινε μια γενική αναφορά για το πώς μπορούν να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια θετική αξιολόγηση τη τάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν προσπάθησε να αναζητήσει λύσει και να εντοπίσει τα μεγάλα προβλήματα. Όμω υπάρχουν δύο θέματα που δεν έχουμε επιλύσει και που είναι συνυπεύθυνα τα κράτη γι' αυτά. Η πολιτική ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η έλλειψη ευρωπαϊκού οικοδομήματος σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στου στόχου και δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα και επίση και η έλλειψη προπολογισμού. Εδώ ακούσαμε την εκπρόσωπο των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα COSME έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια και αυτό εξαρτάται και από τις δημοσιονομικές προοπτικές που το ίδιο το Συμβούλιο περιόρισε σε έναν εφήμερο προϋπολογισμό. Τώρα, ε, μιλάμε γενικά για την απασχόληση, έχουμε 11% και στην Ισπανία βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση, έχουμε φτάσει στο 27% ανεργίας, αλλά δεν μιλάμε για την ποιότητα. Υπάρχουν δύο κριτήρια πάρα πολύ σημαντικά από τη σκοπιά των μικρών και μισών επιχειρήσεων και αυτό είναι η ανταγωνιστικότητα και η αηφορία. Η ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε κόστος. Το κόστος μειώνεται ε, αν μειωθεί το κόστος παραγωγής και μάλιστα μετακυλείται και στους μισθούς και έτσι γίνεται ακόμη περισσότερο ακόμη πιο φτωχός ο πληθυσμός. Ε, κάτι που βλέπουμε ως διαφοροποίηση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης είναι ότι στην Νότια Ευρώπη οι επιχειρήσεις πληρούν πολύ περισσότερο για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ε, δεν ε, βλέπουμε το κοινωνικό ε, συμβόλαιο και η μείωση των μισθών δεν οδηγεί σε καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να βασιστούμε σε φουτουριστικά κριτήρια, σε καλή κατάρτιση, στην καιροτομία και στη δυνατότητα Καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Εγώ ήθελα να κάνω μια κριτική για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη συζήτηση. Είναι σημαντικά θέματα αυτά που πρέπει να επιληθούν. Και όπως ε, λέμε ε, στην Ισπανία πρέπει πραγματικά να επιληφθούμε της κατάστασης και να προσπαθήσουμε να παρέχουμε λύση για τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Γεφλοφικά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας είναι παράγον κλειδί ώστε να ξεφύγει η Ευρώπη από την κρίση και να διευκολυνθεί η δημιουργία της συνεργασίας. Και χρειάζονται κατάλληλοι και καινοτόμοι μηχανισμοί γι' αυτό. Επίσης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα και ευθύνη όπου ανήκει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της να εισαγάγει την ε, την νομοθεσία και όπου δεν ανήκει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της να ενθαρρύνει την νομοθεσία που θα διευκόλυνε επιχειρηματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι έξι γραφειοκρατικές διαδικασίες 12 μέρες και 17,3 από το ε, εισόδημα της επιχείρησης ή ενός νεαρού που θα ήθελε να ξεκινήσει μια επιχείρηση καθιστούν την, την ε, εκκίνηση μιας νέας επιχείρησης για ένα νεαρό ε, επιχειρηματία πάρα πολύ δύσκολη. Πώς μπορεί να διακινδυνεύσει, να διαθέσει τόσο χρόνο και χρήμα αλλά και για τον πιο ηλικιωμένο από την Παγκόσμια Τράπεζα μαθαίνουμε ότι η αναλογία των ε, ηλικιωμένων ή των πιο ε, ηλικιωμένων ε, σε σχέση με τους νεαρούς ε, που θεσπίζουν θέσεις εργασίας είναι αντιστροφή. Αλλά ερωτώ τι είδους επαφή έχετε με τις κυβερνήσεις των κρατών, τι είδους ε, ε, φραγμούς έχετε εντοπίσει, φραγμούς που θα μπορούσατε να βοηθήσετε να καταργηθούν. Υπάρχουν προτάσεις για επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους, υπάρχουν ε, προτάσεις για διάθεση περισσότερων πόρων. Πώς θα παρακολουθήσετε την προτινόμενη κατάρτιση πώς θα παρακολουθήσετε τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας θεωρώ ότι δεν κάναμε αυτό που έπρεπε στο παρελθόν. Κατευθύναμε τους νέους υποψήφιους εργαζομένους σε έναν δρόμο που δεν τους οδηγούσε πουθενά. Ερωτώ λοιπόν εάν θεωρείτε ότι οι διατάξεις οι οποίες επιβαρύνουν με πλέον γραφειοκρατικό ε, κόστος της επιχειρήσης και αναφερθήκατε σε τρεις κύριους παράγοντες και το άρθρο 12 της οδηγίας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, υπάρχουν, επιχειρήσεις, υπάρχουν ε, φορείς που εκπροσωπούν υποτιθέτω τους επιχειρηματίες, αλλά δεν μας έχουν εξηγήσει επαρκώς ε, τι σημαίνουν τα άρθρα αυτά, το 12, το 14. Θα μπορούσατε να μας δώσετε στις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και τώρα δίνω το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Παρακαλώ όμως να είστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι, το πολύ τρία λεπτά, ιδάλλως δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Γκουτιέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους. Λοιπόν, κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχήν, Καλό είναι που από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και την αυτοπασχόληση ως μέσο εξόδου της κρίσης, αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ απαιτητικοί για να χαρτογραφήσουμε τις ε, διάφορες ποικιλίε που υπάρχουν στην αυτοπασχόληση και συμπεριλαμβανομένων και των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Γιατί συμβαίνει κάτι σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδίω σε κάποιες ε, χώρες του ψευδούς αυτοπασχολού που είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να δημιουργήσει αυτοαπασχόληση αλλά ε, να αγκάζεται ε, να το πράξει αυτό γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει να εργαστεί και τελικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα έχουμε έναν ε, τομέα με πάρα πολύ υψηλό επίπεδο φτώχειας γιατί και οι μισθοί είναι πάρα πολύ ε, χαμηλή, αλλά και επειδή οι εισφορές είναι πολύ υψηλές. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τις διαφορές που υπάρχουν για τις μικρές επιχειρήσεις. Ε, ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα για τις πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις και ιδίω για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από 250 εργαζομένους και με ανησυχεί πολύ που αναφέρεστε στην ευελιξία. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία τη στιγμή που συνίσταται μια εταιρεία ε, πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία αλλά με ανησυχεί όταν μιλάμε για απορρίθμιση θέλετε να εισαγάγετε εκεί και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί υπάρχει ακριβώς ε, ένα πρόσθετο αποτέλεσμα. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, ή ε, έχουν εργαζομένους οι οποίοι δεν βρίσκουν εργασία βάσει συλλογικών συμβάσεων και χαίρουν τις λιγότερες τις μικρότερες προστασίας. Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία διάβασα ένα άρθρο της προάλλησης ότι πάνω από το 60% των εργαζομένων που πριν από 10 χρόνια καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσει στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, ε, τώρα δεν ε, καλύπτονται πλέον από αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων και ε, για το θέμα ε, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση έχουμε δύο ουσιαστικά στοιχεία. Καταρχήν ε, έχουμε το θέμα των φόρων, τη φορολογική πίεση. Πολλές φορές έχουμε κάποιες πολιτικές που θέλουν να προωθήσουν την αυτοπασχόληση αλλά αφήνουν ε, στο κοινό τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Παραδείγματος χάρη έχουμε κάποιες φορεκτώσεις που ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά αποκλείονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις. Ε, παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, πληρώνουν 10% ε, με ένα συντελεστή 10% μικρότερο από ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό σε σχέση και με την ανταγωνιστικότητα της πολιτικής καινοτομία, κατάρτισης και της διεθνοποίησης. Ευχαριστώ, κύριος Μπενιούν. Sí, Uh, uh, Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μαρκ Χόγεν γιατί αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις ε, πολιτικές ε, ε, που η, επιχείρηση, η κυβέρνηση συνασπισμού επέβαλε στην ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βελτιώσει την απασχόληση. Δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα για άλλα θέματα, για την μαθητεία παραδείγματος χάρη, που δεν θέλουμε να είμαστε ε, πίσω από τη Γερμανία στην, ε, στα ποσοστά αναργίες και μάθαμε από τη Γερμανία ότι ένα καλό σύστημα μαθητείας βοηθάει. Επίσης θα πρέπει να πούμε για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμα ανέργων και ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μακροχρόνια άνεργους να ξαναμπούν στην αγορά ε, εργασίας και να βοηθήσει την απασχολησιμότητα του εργατικού ε, δυναμικού. Ένα άλλο θέμα που είναι αμφιλεγόμενο είτε έχει θετικές και είναι ότι εργατική, ε, η αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι τόσο αυστηρή όσον αφορά ε, τα τα επίπεδα μισθών και είναι λυπηρό το γεγονός ότι το εργατικό δυναμικό έχει υποστεί ε, πλήγματα όσον αφορά τα έσοδά του. από την άλλη πλευρά υπάρχει και το επιχείρημα ότι τουλάχιστον δουλεύει. Και επίσης κάτι άλλο είναι ότι οι επιχειρήσεις που δουλεύουν ε, και μπορούν να τους απασχολήσουν είναι σε καλύτερη θέση για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη όταν έρθει. Και με αυτή την οικονομική ανάπτυξη θα δούμε ότι και τα επίπεδα των μισθών θα αυξάνονται και θα επωφεληθούν περισσότερο και οι, εργαζόμενοι. Τώρα για τον κύριο Νέμες, αν το λένε έτσι τέλος πάντων. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία λέτε για, την, για τα μυαλά, αν θέλετε, την απορρόφηση μυαλών από τις στοχότερες ε, χώρες στις πλουσιότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό είναι κάπου λογικό, δηλαδή δεν μπορεί να έχει τα ίδια επίπεδο τιμών, ε, το ίδιο επίπεδο αμοιβών σε χώρες με χαμηλό ΑΕΠ σε σχέση με τις χώρες με υψηλό ΑΕΠ. Τα άτομα αυτά, τα μυαλά αυτά μετακινούνται με δική τους θέληση. Ξέρω πολλά πολλά άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο που ήρθαν και έχουν πολλές ε, που έχουν υψηλά προσόντα, είναι ε, εξειδικευμένοι, ε, ήρθανε, δουλεύουν εκεί σε μάσα, αλλά προφανώς σε θέσεις που απαιτούν πολύ χαμηλότερα προσόντα. Από την άλλη πλευρά τουλάχιστον δουλεύουν. Επίσης, για την κυρία Βολζίνσκι θα ήθελα να μας πει λίγα πράγματα παραπάνω για, την, για τις επιπτώσεις, τις αρνητικές επιπτώσεις της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και την ευελιξία στις αγορές εργασίας. Ευχαριστώ σε Σαΐτ Κεμάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, Υπουργό και τους άλλους ομιλητές. Ένα πράγμα ή μια ερώτηση ήθελα να κάνω είναι ε, και από τη, στην αριστερή και, στην, ε, και από την αριστερά, αριστερά και την δεξιά λέμε τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να κάνουν τα κράτη, τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, κοιτάμε το θέμα από πάνω. Από κάτω όμως, η βάση, τι μπορεί να, να γίνει Ξέρω ότι δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να δημιουργήσει κάποιος μια επιχείρηση. Είπε ο υπουργό ένα ε, παράδειγμα. Υπάρχουν όμως και άλλα παραδείγματα. Μια κυρία που είχε έρθει εδώ, η οποία ήταν ε, μεγάλη, την είχε καταλήψει ο άντρας της, μεγάλωσε τα παιδιά της, μεγάλωνε τα παιδιά της ε, μόνη της και ξεκίνησε μια δουλειά με 10, με 10 ευρώ και τώρα έχει εργοστάσιο με 65 άτομα που απασχολεί. Τέλος πάντων υπάρχουν τέτοια παραδείγματα ή δύο νεαροί που δανείστηκαν 50 50 λίρες από τη μητέρα τους για να αγοράσουν ύφασμα, μετά δανειστήκανε την ραπτομηχανή της μάνας τους και ξεκίνησαν μια ολόκληρη επιχείρηση. Ωραία είναι βέβαια είναι αυτά, αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν. Υπάρχουν κέντρα επιχειρηματικής δραστηριότητες, είτε σε... Πολλές φορές βέβαια είναι ανεπίσημη οικονομία ή και μαύρη αγορά τελείως. Όμως οι πολιτικοί πρέπει να είναι πιο ταπεινοί και να δούνε να, να, να, να, σκύψουν λίγο το κεφάλι και να δούνε τι μπορούμε να κάνουν και τι μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να ξεκινήσουν. Υπάρχουν, υπάρχουν ε, διάφορες πρωτοβουλίες, ας πούμε το crowdfunding που γίνεται τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς, δηλαδή ο κάθε καθένας μας μπορεί να ε, βοηθήσει κάποιον να ε, ξεκινήσει μια επιχείρηση. και υπάρχουν και οι μικρο, υπάρχει το microfinancing, η μικροχρηματοδότηση που ε, προσφέρει ευκαιρίες. Τέλος πάντων, θα πρέπει όμως να, μπορέσει να, να μπορέσουμε να επιλέξουμε και τις δραστηριότητες και τα διάφορα project. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα και μπορούν να βρεθούν. Το, το πρόβλημα είναι πώς θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι που θα εξασφαλίσουν μια χρηματοδότηση να μπορούν να προχωρήσουν. Γι' αυτό ακριβώς και η Επιτροπή μας δεσμεύεται να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το microcredit. Ο κύριος Σάρικας, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πάντοτε όταν ζητάτε να μην έχουμε υπερβολική ρύθμιση, όμως θέλω να προσθέσω κάτι ε, να καταργήσουμε τις άχρηστες ρυθμίσεις, ε, όχι τις χρήσιμες. Ε, Παίρνουμε το σκάρι, πρώτη ρύθμιση στην Ευρώπη απαγόρευε να εργάζονται τα παιδιά, οι εγγύες γυναίκες και υπήρχε νομοθεσία για την ασφάλεια των συνθήκων εργασίας έτσι ώστε να υπάρχει προστασία των εργαζομένων, να μην εργαζονται σε κάτεργα. Και εσείς τώρα μιλάτε για την κατάργηση ιστορικών διαδικασιών όπου έχουμε τη βασική προστασία τη ποιότητα ζωή των εργαζομένων, δεν μπορούμε να το προσωπογράψουμε αυτό. Και θέλω να κάνω τρει ερωτήσει στον κύριο Υπουργό. Μιλάμε για την εργασία και οποιοδήποτε θέμα είναι εργασία. Μιλάμε για την αξιοπρεπή εργασία, γιατί υπάρχουν και μη αξιοπρεπεί ε, ε, εργασίε. Δηλαδή, κάποιο που εργάζεται από καθεστώ κλαδιά ε, δεν θα λαμβανόταν υπόψη. Τώρα, σε σχέση με το χρόνο εργασία, έχουμε και άλλο πρόβλημα μαζί σα. Όχι μόνο με τα εκατομμύρια εργαζομένου Βρετανού που επειδή εργάζονται τόσε πολλέ ώρε δεν μπορούν να έχουν προσωπική ζωή, αλλά τώρα έχουμε και πολλούς ε, Βρετανούς εργαζομένους που εργαζόνται με συμβάσεις μηδέν ωρών, δηλαδή είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων 24 ώρες το 24ωρο που να τους καλέσουν να μην τους καλέσουν και δεν ε, χαίρουν ε, δικαιωμάτων όπως είναι η συνταξιοδότηση, η άδεια κτλ. Είναι ουσιαστικά συμβάσεις σκλαβιάς και Ουσιαστικά εγώ έχω κάποια στοιχεία που τριπλασιάζει αυτά που είπατε εσείς. Ε, έχουμε ένα Ινστιτούτο που δίνει τρεις φορές μεγαλύτερο αριθμό από όσα είπε ο Πρωθυπουργό Κάμερον. Πόσος, πόσοι άνθρωποι όμως εργάζονται υπό τέτοιες συνθήκες σκλαβιάς. Και επίσης δύο σχόλια, κύριε Υπουργέ, για αυτό το ίδιο ζήτημα της αξιοπρέπους εργασίας. Σύμφωνα με τα νούμερα που έχουμε εδώ, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει ε, να μειώνεται ε, οι εργαζόμενοι ε, με ε, 8% έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ανέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με ε, την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας τα νούμερα είναι τα διπλά από αυτά που δίνει η δική σας κυβέρνηση και τελικά ποια νούμερα πρέπει να πιστέψουμε, τις δω ή τα δικά σας. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας Μαν. Και θα πω και εγώ δύο λόγια πριν να ξαναδώσω το λόγο στην συγκήτρια. Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Πάντα λέμε το μικρό πάει μπροστά. Χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, με λίγα μέσα μπορούν να προχωρήσουν, κάποιες απλώς χρειάζονται μια διευκόλυνση και μπορούμε να δούμε πολύ ουσιαστικές αλλαγές. Υπάρχουν στην Ευρώπη τέτοιου είδους ευκαιρίες και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και πάνω απ' όλα να ενθαρρύνουμε τον επιχειρηματία για να ιδρύσει μια μικρή ε, ή μεσαία επιχείρηση. Πρέπει να τους ε, πούμε λοιπόν, ναι, μπορείτε να δράσετε, αλλά βέβαια και σε ένα πλαίσιο ε, το οποίο θα είναι πρόσφορο. Έχω, είχα την ευκαιρία να μελετήσω αρκετά το πώς μπορεί μια επιχείρηση να βρει ένα πεδίο πρόσφορο και να λειτουργήσει και να, να ιδρυθεί η εταιρεία από τον επιχειρηματία ο οποίος θα πει ότι να θέλω και να ε, προσλάβω ε, μάλλον ε, νέους ή μάλλον ηλικιωμένους. Δεν πρέπει να λησμονούμε λοιπόν όταν μιλούμε για την απασχόληση των νέων ότι και οι ηλικιωμένοι μπορούν να προσφέρουν ε, πολύ τιμή βοήθεια ε, την εμπειρία που διαθέτουν. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο, παρα... στο περιθώριο και πρέπει να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να εργαστούν και, αυτά, και αυτοί. Δεν αρκεί όμως να μιλάμε μόνο για απασχόληση. Δεν θέλουμε αλλαγή στην, στις στατιστικές. Θέλουμε μια ουσιαστική μεταβολή Άρα χρειάζεται επένδυση στην ποιότητα και όταν λέω ότι η υψηλή ποιότητα που διαθέτουμε στις χώρες μας, η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να δούμε, αποτελεί εμπόδιο για την ε, ένταξη στην επιχειρηματική, για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μπορεί να στηρίξει ακόμη περισσότερο, μπορεί να δώσει ποιοτικέ ε, γνώσεις, κατάρτιση, ευκαιρίες για την ανάπτυξη ε, μιας επιχείρηση την οποία μπορεί κάποιος να μην είχε καν φανταστεί. Αυτό αποτελεί την ποιοτική, αυτό συνιστά την ποιοτική υποστήριξη μπορούμε να προσφέρουμε. Και τελευταία παρατήρηση, θα ήθελα να ξεφύγουμε πλέον από τα λόγια και από το, ε, το ε, χωρίς ουσία, από τις χωρίς ουσία διακήρυξης. Πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε ότι αν κάποιος ε, προσπαθεί να ε, παραβιάσει τους, ε, τις βασικές αρχές και τους κανόνες για την απασχόληση, θα πρέπει να του δείξουμε ότι δρά αντικοινωνικά, ότι είναι βάρος στην ε, κοινωνία και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε για τη δημιουργία των θέσεων εργασία. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, θα ήθελα και εγώ να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που σας φαίνεται, γιατί εγώ βλέπω ότι μάλλον ε, αποδιαρθρώνει την κοινωνική πολιτική με επιχείρημα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ε, αποδιαρθρώνει, διαλύει τελείως το κοινωνικό πλέγμα. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι ένας εργαζόμενος με σωστή ε, προστασία παραμένει ανταγωνιστικός. Είναι ανταγωνιστικός και δεν μπορεί να θεωρείται απειλούμενη η ανταγωνιστικότητα από την, το υψηλό επίπεδο κοινωνική προστασία του εργαζομένου. Από την άλλη για το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελα να επισημάνω ότι όλο το καλοκαίρι βλέπαμε στη, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ε, την ε, συζήτηση αυτή για συμβάσεις με μηδενικές ώρες απασχόλησης. Ε, θα θέλατε να μας πείτε ακριβώς τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η κατάσταση. Τώρα δυστυχώς έχω μόνο ένα 15 λεπτό να σας μοιράσω για να ακούσουμε όλες σας τις ερωτήσεις. Είμαι βεβαία ότι και οι διερμηνείς θα δείξουν την ανοχή με 2-3 λεπτά επιπλέον και άρα ο καθένας σας μπορεί να μιλήσει από 5 λεπτά αλλά με απόλυτη αυστηρότητα ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Κύριε Υπουργέ, εσείς μπορείτε να επιλέξετε σε ποιες ερωτήσεις θα απαντήσετε. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο μέσα στα 5 λεπτά. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και συναρπαστικέ οι παρεμβάσει. Για τον ανταγωνισμό θα ήθελα να πω το εξή, ότι δεν μιλάμε για ανταγωνισμό μόνο μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, αλλά μιλούμε για ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών κρατών. Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο δρόμο. Εάν δεν ε, σταθούμε ανταγωνιστικοί θα χάσει τις εργασίες η Ευρώπη, θα χάσει την ευημερία της και τις, ευ... τις ευκαιρίες για τους νέους. Ε, ας μην μιλάμε μόνο για ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών, να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε και τι συμβαίνει έξω από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, ας ξεπεράσουμε αυτόν τον ε, αποκλεισμό και την Ευρώπη ως... Ε, φρούριο που μας κάνει να λησμονούμε την πραγματικότητα στο οικονομικό πεδίο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι ξεπεράσαμε το, τα προβλήματα στην ε, απασχόληση και τις κακές συνθήκες απασχόλησης των 19ου αιώνα και εισαγαγάμε τις έννοιες της υγείας και της ε, ασφάλειας. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι είχαμε 80 σελίδες με κανόνες για οποιονδήποτε νεαρό ε, επρόκειτο να προσληφθεί σε επιχείρηση με αποτέλεσμα να μην ξέρουν ούτε καν τι σημαίνει δουλειά οι νέοι μας, γιατί δεν τους προσλαμβάνε κανένας. Αυτό ήταν ένα ευρύτατο πλέγμα από νομοθετικές ε, διατάξεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας. Λοιπόν, αυτές 80 σελίδες κάναμε 5 χωρίς να αλλάξουμε το επίπεδο της προστασίας, παραμένουν ενισχύ δηλαδή διατάξει. διατάξεις, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να περιοριστεί η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων. Ο κύριος Μπένιον επίσης μίλησε για τη μαθητεία. Μπορούμε να έχουμε εκατομμύρια ε, θέσεις μαθητείας. Ε, όταν ήμουν εγώ μικρός, ε, μαθητεία προσέφεραν τα ορυχεία, τα ναυπηγεία, ενώ τώρα μπορούμε να έχουμε στην παροχή φροντίδα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση, θέσεις μαθητείας λοιπόν, στάζ, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να επενδύσουμε στους νέους, να βοηθήσουμε την παραγωγικότητά τους, να βελτιώσουμε το δυναμικό τους και να τους επιτρέψουμε να είναι ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια αγορά. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν με την κατάρτιση αυτού του τύπου, με τη μαθητεία και επίσης ή την ε, πρακτική άσκηση. Επίσης... Ε, μπορούμε και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζει σαν, ενδεχόμενο η, σαν ενδεχόμενη λύση η Ισπανία αυτή τη στιγμή για να καταπολεμήσει την ενεργεία της. Δίναμε επιδοτήσεις σε εργοδότες εφόσον μπορούσαν αυτοί να προσλάβουν και να δώσουν μια ευκαιρία για την αγορά εργασίας κάποιων ε, μακροχρόνια ανέργων για την ε, καταναγκαστική εργασία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι σημαίνει αυτό. Η ανελαστικότητα στην αγορά εργασίας πολλές φορές μπορεί να αποτελέσει παράγοντα για καταναγκαστική εργασία. Η ανελαστικότητα φέρει πριν στην τελική αγορά εργασίας από ό,τι μου λένε πολλοί συνάδελφοι από την Ιταλία. Είναι αυτή η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και εντείνεται ο κίνδυνο της ανεργίας για τις ε, συνθήκες διαβίωσης και τις ε, συμβάσει εργασίας με μηδενικές ώρες έργου. Ε, θα ήθελα να σα πω το εξή, ότι η αύξηση στην απασχόληση το τελευταίο χρόνο στο Ρωμανό Βασίλειο είναι μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση. Αυτά είναι στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Όταν κανείς εργάζεται σε πλήρους όρους απασχόλησης, ε, σε πλήρου όρου απασχόληση δεν μπορεί να καταγραφεί ως άνεργος και με μόνιμη θέση εργασία. Αυτά είναι τα στοιχεία της ε, ILO ε, και πρόκειται για τάση αντίστροφη από αυτή που είχαμε δει ε, πριν από την κρίση. Θα ήθελα να πω βεβαίως ότι αυτό το προσφέρει σαν ευκαιρία η ευελιξία γιατί μπορεί κάποιος εργαζόμενος να θέλει να μπορεί να ρυθμίσει πόσες ώρες θα δουλεύει ή ποιες ώρες θα δουλεύει ώστε να τη συνδυάσει και με την οικογενειακή ή προσωπική του ζωή. Ε, τώρα, το, αυτή, η δυσμενής εικόνα που δόθηκε για τις ε, συμβάσεις εργασίας με μηδενικές ώρες απασχόλησης είναι απλώς μια κακή εικόνα που προβλήθηκε εις βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου για να δυσφημιστεί. Πρέπει να σας πω ότι εάν δεν υπάρχουν δυνατότητες της ευελιξίας, να, ε, δεν θα μπορεί ο εργοδότης να προσλαμβάνει εργαζομένους. Ας μην Ας μην παραγνωρίζουμε λοιπόν την αξία και ας μην δείχνουμε ασέβεια απέναντι στην ε, περιορισμένη επασχόληση, στη μερική επασχόληση γιατί αυτή μπορεί να δίνει ευκαιρία για μετάβαση σε μια πιο μόνιμη θέση εργασία αργότερα. Και ας κοιτάξουμε και πριν από την κρίση τι συνέβαινε, ότι μπορούσαν αυτοί που εργάζονταν να έχουν αυξήσει στις τάξεις του 10-15%, να έχουν και τη σχετική κοινωνική πρόνοια κτλ. Ενώ οι λοιποί βρίσκονταν εξαρτώμενοι από ένα επίδομα ε, ανεργία. Ε, τώρα ο προτιμάει, αντί να δει την αύξηση στο, δικό του μισθό, να ξέρει ότι και τα παιδιά του και τα εγγόνια του θα έχουν μία θέση εργασίας. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε για να κλείνω είναι να έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά, να επενδύσουμε στους ανθρώπους, να έχουμε μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας, να επενδύσουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία και αυτό να σημαίνει ότι επενδύουμε στο, στην καλύτερη οικονομία και στο καλύτερο εργατικό δυναμικό του κόσμου. Διαφορετικά θα δούμε και πιο πολλούς ανέργους και πιο πολύ ακόμη υποβάθμιση των συνθήκων διαβίωσης. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα δώσω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρο μας Μάν, αλλά να δώσω το λόγο και στον κύριο Νιμίκα και λυπάμαι που δεν θα μπορούσα να ακούσω την απάντησή του. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε τρία σημεία γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να απαντήσω σε όλα όσα ακούστηκαν. Καταρχήν, για το θέμα της ρύθμισης. Θα πρέπει να δούμε το ζήτημα σε πιο ευρύ πλαίσιο. Εμείς ε, επιμένουμε σε θέματα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας ε, και συχνά μιλάμε για τομείς ρυθισμένους με υψηλή προστασία οργαζομένων. Ε, Αυτή η τομή είναι η πιο ανταγωνιστική. Αυτό συμβαίνει κυρίως στη βιομηχανία και αν δούμε ποιες, χώρε χώρες σημειώνεται τέτοια επιτυχία, στις σκανδιναβικές χώρες αλλά και στη Γερμανία, στο βιομηχανικό τομέα όπου υπάρχουν υψηλά πρότυπα, όχι στις υπηρεσίες. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αν θέλουμε ανταγωνιστικές και κοινοτόμες επιχειρήσεις. Και πολύ συχνά αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν να ε, καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες ε, οι επιχειρήσεις για την καινοτομία περισσότερο παρά για το κόστος εργασίας, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Και ξέρω από τις συζητήσεις ε, που είχα με τα κράτη-μέλη, τα οποία μπήκαν ε, πιο μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πολύ συχνά αυτά τα κράτη στοιχημάτισαν και επένδυσαν στην ανταγωνιστικότητα, όμως ε, αυτά τα, τα ποινικοποίησε και θα τα ποινικοποίησε και στο μέλλον. Ε, και πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση στα άτομα και στην κοινοτομία και στην έρευνα. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε και τα κατάλληλα μέσα. Νομίζω ότι αυτό είναι το συμφέρον μας. Τώρα, αυτό συνδέεται και με το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής. Πράγματι, θα θέλαμε μια πιο ενεργητική προσέγγιση για το ζήτημα αυτό, γιατί κατανοούμε ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα στοιχεία εξέλιξης και ελπίζω ότι θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με τους εργοδότες. Δεν θα δούμε μόνο την εφαρμογή των κανόνων εσωτερικής αγοράς. Έχουν εφαρμοστεί αυτές οι νομοθεσίες κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα και είδαμε που μας οδήγησε αυτό όμως σε ορισμένου τομεί όπου προωθήσαμε τη συνεργασία είδαμε να στεφτεί με επιτυχία η δημιουργία θέσεων εργασία στην ΕΡΒΑΣ παραδείγματο χάρη, γιατί δεν προσπαθούμε να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση περισσότερο Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη πολιτική ολοκλήρωση και προσπάθειες σε ορισμένους τομείς, ε, αλλά και κάποιες ε, συνθήκε ε, πρέπει να ισχύουν. Παίρνουμε το χάρη στον τομέα τη ενέργεια. μπορούμε να έχουμε κέρδη παραγωγικότητας και να έχουμε και χαμηλότερε δαπάνες αν συνεργαστούμε. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το ποιο τρόπο εξελίσσεται ο ανταγωνισμός ανάπτυξης του υπόλοιπου κόσμου. Καταρχήν, τι βλέπουμε. Η κρίση και η οικονομική διακυβέρνηση οδήγησαν στον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών ε, για την ε, μείωση των μισθών, η μισθή προς τα κάτω. Γιατί αυτό που έχει επιβληθεί από για την Νότια Ευρώπη είναι η μείωση των μισθών ε, πέρα από την εξυγίανση ε, των δημοσιονομικών και αν, ε, αν ακολουθήσουμε αυτή την οδό μπαίνουμε σε ένα κύκλο. γιατί βλέπουμε τι έγινε στην Ελλάδα, στην Ισπανία, αλλά θα είναι η Γαλλία η επόμενη χώρα που θα τεθεί υπό επίθεση και αν υποχωρήσει η Γαλλία θα βρεθεί σε προβληματική κατάσταση και η Γερμανία και Πρέπει να δούμε και τις συνέπειες. Οι συνέπειες είναι ότι ε, δυστυχώς χάνουμε θέσεις εργασίας, χάνουμε εισοδήματα. Μιλώ για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και αμφισβητείται εδώ η εμπιστοσύνη των εργαζομένων διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων Και δεν βλέπουμε δυστυχώ ε, πολύ μεγάλη αντίθεση αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό project, αλλά θα μπορούσε να γίνει. Εγώ είχα μια μικρή εμπειρία στην Πολωνία για ένα project που πολιτικά παρουσιάστηκε από του κομμουνιστές και υποτίθεται ότι θα, προσ... θα χάριζε ευτυχία σε όλου, αλλά τελικά απορρίφθηκε. Αν οργανώσουμε λοιπόν τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσχόμενοι περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά μείωση, αλλά μάλλον με ε, κόστος να έχουμε τη μεγαλύτερη επισφάλεια, αυτό συμβαίνει σήμερα. Και το τρίτο πολύ σύντομο στοιχείο, για να απαντήσω στην κυρία Σλοβέσκα. Ναι, ε, προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτό. Το εγχείρημα της ανάλυσης της αγοράς εργασίας αποτελεί στοιχείο αυτής της προσπάθειας, αλλά ταυτόχρονα ταυτόχρονα δεν, γίνεται, δεν ακολουθείται η σε εθνικό επίπεδο. Στην Πολωνία, παραδείγματο χάρη, μα ενημέρωσαν συνάδελφοι ότι με του Πολωνού προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο, όμω δεν στεφθεί με επιτυχία. Ίσως ε, τώρα να ξεκινήσουν μια νέα προσπάθεια και θα δούμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλώ την ε, κυρία Βοροζίσκη να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά, αν δεν έχετε αντίρρηση όμως. Μια και είμαι η τελευταία ομιλήτρια, θα είμαι σύντομη. Κυρία Γιαζεύσκα, μιλήσατε για το monitoring, κυρίως όσον αφορά την δημιουργία των επιχειρήσεων από τους νέους. Αυτή είναι, αυτός είναι από τους βασικούς στόχους του Small Business Act και αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει σε συνεργασία όπου θα εξετάσουμε μάλλον όλα τα θέματα της ταχύτητας, της ευκολίας, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από τα μοντέλα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Το monitoring όσον αφορά την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους και φαντάζομαι δεν μιλάτε για την αρχική επένδυση αλλά και για την ε, συνεχή κατάρτιση. Αυτό είναι ένα ένας από τους βασικούς μας ε, στόχους, όμως θέλουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να το κάνουμε σωστά και στηριζόμαστε στην ικανότητα των μελών μας. Και για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό, γιατί είναι ένα θέμα ε, της, ε, ε, ε επιστροφής, της της επένδυσης. Ε, και κυρίως η απόσπαση για το άρθρο 12 θα να, κάνουμε, να έχουμε ένα ραντεβού για να σας εξηγήσω διμερώς ε, αυτό το θέμα της ε, κοινή ευθύνη θα δημιουργήσει προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν υπεργολαβίες γιατί θα, θα υπάρχουν και προβλήματα με τις αρχές των θα πρέπει να κάνουν τους ελέγχους, δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντικαθιστήσουν, αντικαθιστούν στις αρχές. Τώρα κύριε Πριέτο, ε, αυτό που, γι' αυτό που είπατε είναι πραγματικό, μένα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να τα να, να, να, να, λειτουργήσουμε ε, αυθαίρετα. Ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ε, για τον κύριο Μάνα, για την μη δηλωμένη εργασία. Είμαστε υπέρ της καταπολέμησης της μη δηλωμένη εργασίας. Μας συμμετέχουμε σε μια διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κοινωνικούς εταίρους, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η μη δηλωμένη εργασία είναι εις βάρος των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, το θέμα της, ε, του κανονισμού για τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Ποιο είναι το πιο χρήσιμο. Ναι, συμφωνούμε, αλλά για το ε, για την άσκηση refit που έθεσε και η πρόεδρος. Θα πρέπει να δούμε πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι δυσανάλογη για τις, όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς δεν θέλουμε μία νομοθεσία, θέλουμε έναν κανονισμό ο οποίος να είναι καλύτερα προσαρμοσμένος στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ και για την κατανόηση. Και πάλι τα τελευταία τελευταία λόγια στην ε, κυρία, η συγγήτρια. Δύο λεπτά, αλλά όχι περισσότερο. Thank you very much. Well, really, I want to thank... Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις προσκεκλημένους μας που ήρθαν εδώ και μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας και κυρίως τον κύριο Χόμπαν γιατί δεν έχουμε πολύ συχνά έναν υπουργό που να θέλει να έρθει να στην Επιτροπή μας. Επίσης ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους ε, που ε, έκαναν πάρα πολλά σχόλια, πολύ ενδιαφέροντα τώρα. Εγώ ε, συγκράτησα δύο τεινά Κάτι που ακούστηκε πολύ είναι το θέμα της ε, μείωσης ε, της νομοθεσίας της απορρίθμισης και ασχοληθήκαμε και με το θέμα της νομοθεσίας ε, για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο Το θέμα είναι να προβούμε στην μείωση τη νομοθεσία χωρί να μειώσουμε την προστασία των εργαζομένων και του εργατικού δυναμικού. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι πολύ καλό ότι ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και ακούσαμε κάποια παραδείγματα σήμερα. Επίσης, ε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα την εμπειρία της κυρίας Γεροβλέσκα σε σχέση με ε, την ίδρυση μιας επιχείρησης που πρέπει να αντιμετωπίσει έξι διαφορετικές διαδικασίες μέσα σε ένα μήνα. Αν μπορούμε να το περιορίσουμε, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Και το θέμα της σημασίας της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας ε, από το σχολείο και μετά. Το Πανεπιστήμιο για την δική μου περιοχή άνοιξε ε, τα γραφεία του εδώ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα αποκαλούνται το Πανεπιστήμιο των Ευκαιριών και το 75% των φοιτητών ε, το παίρνουν από την ε, περιοχή των μαύρων και το 90% των αποφύτων του πανεπιστημίου αυτό βρίσκουν δουλειά. από την περιοχή των ορυχείων. Έτσι λοιπόν παίρνουν τους φοιτητές τους. Θα προσπαθήσω πάντως να τα συμπεριλάβω όλα αυτά μέσα στην περιορισμένη εκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για την κατανόηση, για τη συντομία, για τις ε, πολυδατικές ανταλλαγές απόψεων. Ιδιαίτερος ευχαριστώ όλους τους εδώ παρόντες και τους ερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ξεπεράσαμε κάπως το χρόνο μας. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.